Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ε, ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες της Επιτροπής μας με την ημερήσια διάταξη που είναι πάρα πολύ πλούσια ε, γιατί επανερχόμαστε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές με μια πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη και τα πιο σημαντικά θέματα της ημερήσιας ε, διάταξης είναι η προστασία των ζώων, ε, η βία που ασκείται έναντι των ζώων. Πάρα πολλοί πολίτες και από διάφορα μέρη της Ευρώπης απευθύνθηκαν στην Επιτροπή μας και έφτιαξαν το θέμα αυτό. Μετά έχουμε μια μια αίτηση σχετικά με τα περιβαλλοντικά στη Μεγάλη Βρετανία και θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση ε, για το τι έγινε στην Δανία και σε άλλες χώρες κατά τους προηγούμενους μήνες. Θα έχουμε και την ψηφοφορία για την ετήσια ε, έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής μας του 2012. Ο κ. Μακμίλαν Σκοτ θα παρουσιάσει το θέμα αυτό και επίσης έχουμε και την άποψη του κ. Τσίτσεστερ σχετικά με, τις, ε, με τη δυνατότητα που υπάρχει να ε, διατηρηθούν οι δύο έδρες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατόπιν θα υπάρξει και μια συζήτηση για τις αναφορές που έχουν καταθέσει αρκετοί σχετικά με την υλοποίηση Notre Dame de Londres. Επίση, ε, θα υπάρχουν και εκπρόσωποι από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλον, όπω και οι αναφέροντε που κατέθεσαν τι μεμονωμένε αναφορέ. Η ημερήσια διάταξη ε, προβλέπει και την ε, ψηφοφορία, όπως σας είπα, αύριο το πρωί, για να μην υπάρχουν λοιπόν τα προβλήματα. Το πρώτο σημείο που είναι ανακοινώσεις του Πρόεδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών θα προηγηθεί αυτό. Οι ψηφορίε θα ξεκινήσουν στις 9 και 4 και πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 10. Και αυτό θα το προσπαθήσουμε να το συνδυάσουμε με ένα επίσημο αίτημα που κατατέθηκε από μία σειρά συναδέλφων, οι οποίοι επιθυμούν το θέμα σχετικά με την ψηφοφορία της έκθεσης σχετικά με την αποστολή στη Μαδρίτη, αυτό να ψηφιστεί αμέσως μετά τις δύο εκθέσεις, τις οποίες έχουμε ήδη εντάξει για ψηφοφορία στην ημερήσια διάταξη. Όπως σας είπα λοιπόν, θα έχουμε εδώ εκπροσώπους ε, της γαλλικής πλευράς σχετικά με το Notre Dame de Land. Ε, έχουν κατατεθεί αναφορές σχετικά με το θέμα αυτό και σήμερα θα ξεκινήσουμε με την αναφορά σχετικά με την κακομεταχείριση και την προστασία των ζώων. Και για κάθε μία αναφορά έχουμε παρόντα και έναν από τους ε, αναφέροντες. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Και νομίζω ότι αυτά είχα να σας πω σχετικά με τη Μισελ. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο σημείο και στο δεύτερο αυτό σημείο της ημερήσιας διάταξης έχουμε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 24 μέχρι 25 Απριλίου, 27 με 28 Μαΐου, 19 Ιουνίου και 8 με 9 Ιουλίου. Είναι τα πρακτικά τα οποία έχουν δημοσιευτεί και κατόπιν τούτου νομίζω ότι όλοι σας μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα πρακτικά. Ε, κατόπιν τούτου ε, εγκρίνονται τα πρακτικά, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, άρα εγκρίνονται τα πρακτικά. Πάμε στο τρίτο σημείο. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Θεωρώ ότι πρέπει ε, να ε, καλωσορίσω επίσημα την Ρίντα, η οποία ασχολήθηκε με πάρα πολλά θέματα, τα οποία είναι σημαντικά κυρίως ε, σε σχέση με τις ισπανικές αναφορές και την ε, ανακάλυψαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που προσέφερε μέχρι σήμερα στην Επιτροπή μας και της ευχόμαστε καλή δουλειά για, τις, ε, τη μελλοντική της εργασία. Ε, να καλωσορίσω και την Ναταλία Παπαστεριάδου, η οποία ήρθε και αυτή στο δικό μας το οργανόγραμμα. Δεν τη βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει την καλωσορίζω στην οικογένειά μας, στην Επιτροπή των Αναφορών. Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις. Κατόπιν τούτου, αν δεν επιθυμεί κάποιος να λάβει το λόγο, θα ήθελα να περάσουμε ευθύ αμέσω στην ημερήσια διάταξη. Και όπως σας είπα, ξεκινάμε με τη συζήτηση σχετικά με τα θέματα που έχουν σχέση με τα ζώα. Ξεκινώ λοιπόν με την 595 του 12 μια αναφορά την οποία θα παρουσιάσει η συνάδελφος κυρία Μουσκαρντίνη, την οποία και καλωσορίζω. Έχει υπογραφεί αυτή η αναφορά από 349 αναφέροντες και αυτή η έκθεση ε, κατατίθεται εκ μέρους ε, των Ιταλών οι οποίοι τίθενται κατά της ζωοτομίας και κατά της ε, κτηνοβασίας με τα ζώα. Έχετε λοιπόν το λόγο για να μας παρουσιάσετε την αναφορά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως θα θυμάστε, στην συνεδρίασή μας είχαμε διάφορες αναφορές που αφορούν ε, στην κακομεταχείριση των ζώων. Και νομίζω ότι ένα από τα ε, νέα προβλήματα θα έλεγα σε σχέση με το παρελθόν είναι το θέμα της ε, σεξουαλικής ε, επαφής με τα ζώα. Κτηνοβασία δηλαδή, η οποία υπάρχει δυστυχώς σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχουν βέβαια και νομοθεσία, υπάρχει και νομοθεσία που απογορεύει κάτι τέτοιο, όπως στη Γερμανία, ενώ στην Ιταλία δεν προβλέπεται ακόμα τέτοιου είδους νομοθεσία και απαγόρευση. Και έχουμε και άλλες χώρες που όπως απορρέει από τα έγγραφα τα οποία έχουμε αποστείλει στην Επιτροπή μαζί με την αναφορά, από αυτά τα έγγραφα απορρέει, όπως τη Δανία ας πούμε, Υπάρχουν ε, χώροι μάλιστα όπου ε, με αμοιβή πληρώντας μπορεί κανείς να έχει σεξουαλική επαφή με τα ζώα. Αυτές λοιπόν ε, είναι ε, αγγελίες ε, που εμφανίζονται και σε εφημερίδες και σε διαδικτυακούς τόπους. Γι' αυτό λοιπόν μαζί με τα έγγραφα που σας έχουμε αποστείλει σας στέλνουμε και πάρα πολλές φωτογραφίες που υπάρχουν τόσο για ακτινοβασία όσο και για κακομεταχείριση όσον αφορά τη ζωοτομία. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι πάρα πολλά πειράματα. Είναι πειράματα ε, που δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι πονάνε τα ζώα για να σωθούν οι άνθρωποι. Κάτι άλλο. Πρόκειται για πειράματα τα οποία είναι περιτά και τα πειράματα αυτά απλά αποφέρουν χρήματα χρήματα σε μεμονωμένες ομάδες, σε πανεπιστήμια ή σε ενώσεις που κάνουν αυτά τα πειράματα και με τον τρόπο αυτό προκαλούν περιττό πόνο σε εμβιόντα όπως είναι τα ζώα. Η Ευρώπη λοιπόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις ε, εκλήθη να τοποθετηθεί, όπως είπαμε το Σχάριν, για την νομοθεσία σχετικά με τη ζωοτομία. Εκεί έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος. Όμως, δυστυχώς, υπολείπονται ακόμα πάρα πολλά και γι' αυτόν το λόγο κατατέθηκε αυτή η αναφορά την οποία έχουν υπογράψει τόσα πολλά άτομα και θα την υπογράψουν και άλλοι. Θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε και εμείς πιστεύουμε ότι η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να καταδικάσει απερίφραστα τα γεγονότα αυτά, να ζητήσει από την Ευρώπη ενιαία νομοθεσία έτσι ώστε να απαγορεύει την κτηνοβασία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ε, ευχαριστούμε κυρία Μουσχαρντίνη, λέει πρόεδρος, και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Λορέντσο Κρότσε, ο οποίος έχει υπογράψει και αυτό στην αναφορά. που δεν ήρθε όμως. Η κυρία Μουσκαρντίνη, νομίζω ότι τον κύριο Κρότσο αντικαθιστά ο δικηγόρος Τσεκών, ο οποίος ε, μπορεί να λάβει το λόγο. Μου λένε ότι δυστυχώς του έτυχε κάτι απρόπτο και έστειλε ένα έγγραφο το οποίο διανεμήθηκε στα μέλη της Επιτροπής from the Commission. Anyone, Mr. Hansen. But we have not anyone else? Not on this one. Not on this item. Next item. Allora, do la parola per la Commissione. Λοιπόν, ε, ο κύριος Χάνσεν έχει το λόγο εκ μέρους της Επιτροπής. Thank you very much. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και εσείς αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Λέγομαι Μπιόν Χάνσεν και είμαι τμήματάρχης της ε, αρμόδιας γενικής διεύθυνσης που είναι και η κυρίως αρμόδια για την οδηγία για τα πειραματόζωα. Είπατε κυρία Πρόεδρε ήδη ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν θα επαναλάβω τα όσα έχουμε περιλάβει στο έγγραφό μας. Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτε άλλο από, σε αυτά δηλαδή που έχουμε ε, ήδη ε, θέσει επί χάρτου και γι' αυτό θα αρκεστώ σε αυτά κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Έχω κάνει την εξή ε, έκκληση στους ε, εκπροσώπους της Επιτροπής για να κερδίζουμε χρόνο να μην επαναλαμβάνουν αυτά που αναφέρονται στα έγγραφα. Αλλά θέλω να επαναλάβω ότι η παρουσία μας ε, εδώ έχει ως νόημα το να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις ε, και γι' αυτό σας δώσαμε το λόγο. Εν πάση περιπτώσει θα δώσω τώρα το λόγο στους ε, συναδέλφους και στην περίπτωση που δεν τοποθετηθεί η Επιτροπή στα θέματα που έχουν τεθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να καταθέσει γραπτά την άποψή της και εκεί να αναφέρεται βέβαια σε όλα τα θέματα που όμως όπως σας είπα μπορεί να μην είναι όλα τα θέματα τα οποία τίθενται στις αναφορές. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψη των συναντέλφων επί του θέματος. Υπάρχει κάποιος παρακαλώ που επιθυμεί να λάβει το λόγο. Η κυρία Χόκεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τα πειράματα με ζώα. έχουν να στη Δανία. Υπήρξα μέλος κυβερνητικής επιτροπής που προέβη στην αξιολόγηση των ε, πειραμάτων σε ζώα και εγώ κατά κάποιο τρόπο ήμουν εκπρόσωπος των ζώων. έχουν να ότι εάν υπάρχει αυστηρή νομοθεσία που θα πρέπει να υπάρχει και στην Ένωση και στον ΩΣΑ και εφόσον τηρείται η νομοθεσία αυτή, τότε έχει καλώς διότι έχουμε θεσπίσει αυστηρούς κανόνες. Όχι μόνο για τα πειράματα, αλλά και, και την φάση εκείνη της ζωής των ζώων μεταξύ πειραμάτων. Να μην είναι δηλαδή χωμένα απλά σε ένα κλουβί. Τώρα όντως, τουλάχιστον θεωρητικά, προστατεύονται καλύτερα τα ζώα σε πολλές από τις χώρες μας. Το ίδιο για τη γεωργία. Ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζονται τα ζώα ε, στην γεωργία είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να μας απασχολεί. Εάν λοιπόν η νομοθεσία που ισχύει για τα πειράματα σε ζώα ε, τηρείται αυστηρά, τότε είναι και υπερβολικά δαπανηρό να κάνει κανείς πειράματα σε ζώα. Τώρα, γνωρίζουμε ότι η βιομηχανία, εν ώψη αυτού του γεγονότος, δεν θέλει πλέον να κάνει πειράματα με ζώα. Αν λοιπόν βρουν εναλλακτικό τρόπο να κάνουν τα πειράματα, θα τον χρησιμοποιήσουν. Πάντα υπάρχουν δύο πλευρές στο ίδιο θέμα. Έχουμε και το νόμο για τα καλλιντικά. Γνωρίζετε ότι έχουμε και πολλή ε, διαφήμιση και μάρκετινγκ ε, στην Ευρώπη για υπερπροϊόντων τα οποία δεν έχουν προκύψει από πειράματα σε ζώα. Αλλά ορισμένες χώρες έχουν αδύναμη νομοθεσία. Τώρα, εάν κάποιος αρρωστήσει λόγω της χρήσης ενός προϊόντος, θα είναι πολύ δύσκολο να ε, αντιμετωπίσει το δικαστήριο με τέτοια περίπτωση. Στην Αμερική βέβαια αν ήσασταν θα έχετε ολόκληρο στρατό δικηγόρων να σας ε, υποστηρίξει την υπόθεσή σας εάν ένα προϊόν δεν είναι ασφαλές. Αυτό θέλω να πω ότι υπάρχουν πάντα δύο πλευρές. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί σε ό,τι αφορά τις συνθήκες για τα πειράματα με ζώα, σε όλη μάλιστα την διαδικασία και Βεβαίω να μην πλανόμεθα όταν λένε ορισμένοι ότι μπορούν να κάνουν τα πράγματα, τα πειράματα αυτά και χωρί ζωά, μπορεί απλά να το κάνουν για λόγους εξοικονόμησης ε, χρημάτων. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε για το θέμα αυτό. Η συνάδελφος κυρία Μουσκαρντίνη, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να επανέλθω, γιατί ξέρετε έχω την εντύπωση ότι για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάλαβε για τι πράγμα συζητάμε. Και αν αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ή προσποιείται ότι δεν κατάλαβε και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Εδώ και χρόνια πολίτες από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βουλευτές, ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες σε διάφορες θητείες καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί ξεκάθαρα σχετικά με την κτηνοβασία, με την παράνομη διακίνηση των ζώων, πάνω στο πρόβλημα των ζώων ε, που ε, χρησιμοποιούνται και εκτρέφονται σε κλουβιά και επίσης Κάτι άλλο που το είπα λίγο πριν είναι ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ε, απαγορεύσει ρητά την κτηνοβασία. Η Κομισιόν προφανώς ε, κερδίζει χρόνο ε, και λέει για να κερδίσει χρόνο στείλτε μας ένα έγγραφο. Αλλά σας λέω υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα και η Κομισιόν σιωπά όπως ε, σιωπά όλα αυτά τα χρόνια που δεν είναι σωστό. Εγώ εκπροσωπώ όλους αυτούς τους πολίτες και ρωτώ την Επιτροπή κατά πόσον προτίθεται να καταθέσει ε, την ε, απαγόρευση σεξουαλικής επαφής ανάμεσα σε ανθρώπους και ζώα. Προτίθεται να το πράξει αυτό η Επιτροπή, ναι ή όχι. Πρόεδρος, νομίζω, μισό λεπτό, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Yes. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να επανέλθω. Είχα πληροφορηθεί ότι έχετε αρκετά επιβαρημένη ημερησία διάταξη και επειδή έχουμε διατυπώσει σαφώς τις θέσεις μας εγγράφως θεώρησα ότι η προηγούμενη παρέμβασή σου μπορούσε, μου μπορούσε να είναι πολύ σύντομη. Γι' αυτό λοιπόν την κράτησε όσο γίνεται συντομότερη. Φαίνεται όμως ότι παρανοήθηκε και γι' αυτό επιθυμώ να απαντήσω στην ερώτηση και επομένως θα καταναλώσω χρόνο και να με συμπαθάτε γι' αυτό, διότι άλλοι ίσως θα έχουν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους μετά. Ορισμένα από τα θέματα που θέτει η αναφορά δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης και είναι καθαρά αποκλειστικής αρμοδιότητας των χωρών μελών, όπως ορισμένα θέματα κτηνοβασίας, καθώς και άλλα τα οποία θέτει η έκθεση. Τα ζητήματα, νομίζω, που εμπίπτουν σε κοινοτική αρμοδιότητα, ενωσιακή αρμοδιότητα, είναι εκείνα που έχουν σχέση με την χρήση ζώων για πειραματικούς σκοπούς, για το χώρο αυτό δηλαδή όπου η Κομισιόν έχει το δικαίωμα υποβολής προτάσεων. Το έχουμε πράξει αυτό με οδηγία η οποία εγκρίθηκε το 2010. Η εν λόγω οδηγία, όπως εξηγούμε στο έγγραφό μας, εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή προστασία για ζώα που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς η νομοθεσία βελτιώνει σημαντικά την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς σε σχέση με την προηγηθήσα οδηγία που χρονολογείται από τα τέλη δεκαετίας του 80 αν θυμάμαι καλά. Επίσης, διοχετεύει περισσότερους πόρους για την αξιολόγηση και ανάπτυξη άλλων εναλλακτικών μεθόδων, κυρίως με την ενίσχυση του ΕΚΒΑΜ, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αξιολόγησης Εναλλακτικών Τρόπων και Μεθόδων που είναι, βρίσκεται στην Ίσπρα της Ιταλίας. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι και ο καλύτερος δρόμος προς τα εμπρός, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε και να αποφύγουμε την χρήση των ζώων για πειραματικούς σκοπούς. Είναι σημαντικό εν προκειμένου όταν μιλούμε για πειραματόζωα και για την χρήση τους για πειραματικούς σκοπούς, να δούμε ότι υπάρχουν δύο πτυχές. Αφενός η ασφάλεια, που έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ασφάλεια και πάλι των προϊόντων που διατίθεται στην ενωσιακή αγορά, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα πειραματόζωα που θα χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στον χώρο αυτό δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια για παράδειγμα ιατρικών συσκευών, προϊόντων, φαρμακευτικών κτλ. με την χρήση μόνο μεθόδων που να μην έχουν ανάγκη από πειραματόζωα παρόλο που θα θέλαμε να υπάρξει τέτοια εξέλιξη. Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει για την ώρα. Άρα επενδύουμε σημαντικά η Κομισιόν δηλαδή στα προγράμματα του ορίζοντος 2020 αλλά και στα πλαίσια των ενεργειών του ε, Κοινού Κέντρου Ερευνών στην ανάπτυξη μεθόδων που θα μας επιτρέψουν να μην χρησιμοποιούμε πειραματόζωα στο, στο μέλλον. Λοιπόν, εδώ είμαστε πολύ δραστήριοι. Έχουμε και την οδηγία και επενδύουμε και σημαντικά. Σε όλους τους άλλους τομείς που αναφέρει η ε, αναφορά δυστυχώς είναι εκτός της αρμοδιότητας της Ένωσης και εμπίπτουν στην επικουρικότητα. Επομένως η Κομισιόν δεν μπορεί να έχει άποψη για το εάν χρειάζεται να αναλυφθεί δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι έτσι και σας εξήγησα την έντονη προσπάθειά μας να μειώσουμε την χρήση των πειραματοζώων, αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι μπόρεσα να σας εξηγήσω και γιατί δεν έχουμε λεπτομερή τουλάχιστον άποψη για θέματα τα οποία εκπίπτουν των αρμοδιοτήτων μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δώσατε αυτό τον έξτρα χρόνο για να εξηγήσω την θέση μας. Ευχαριστώ. Στριφλέρ, δεν ήθελα να παρέμβω, αλλά η απάντηση σας με έκανε να στήσω το λόγο ε, σας μίλησε η συνάδελφός μου για την κτηνοβασία, σας μιλήσατε διαμακρών ε, για τα πειράματα σε ζώα. Ε, εντάξει, αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω τότε, σε τι χρησιμεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δεν ασχολείται με το άρθρο 13 της Συνθήκης Λισαβόνας, ε, αν το γράφει στα παλότερα των υποδημάτων της αυτό το άρθρο. Εγώ πραγματικά ντρέπομαι να, ακούσω, να ακούω τέτοιες απαντήσεις, διότι βλέπουμε να εξαπλώνεται η κτηνοβασία και ντρέπομαι να ακούω τέτοιες ε, απαντήσεις με τόσες υπεκφυγές από την Κομισιόν. Είναι αξιοθρύνητο, λυπούμε πολύ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο κυρία Στρέφλα και εγώ προτείνω να γκρίνουμε αυτά τα οποία ελέγχθησαν για αυτή την αναφορά. Θα ακούσουμε βέβαια και τι ακόμα θα λεχθεί. βάση τόσο σε γενικές γραμμές ε, συμφωνούμε με αυτά ε, που μας είπε η Επιτροπή, η οποία βέβαια είναι αρκετά αυστηρή όσον αφορά την περιχαράκωση των ε, αρμοδιοτήτων της. Πάντως, η ε, ευαισθησία που υπάρχει από αυτή την Επιτροπή νομίζω δεν επιτρέπει να κλείσει το όλο θέμα. Ας παραμείνει λοιπόν ανοιχτή η αναφορά και θα δούμε μετά τι μπορούμε να κάνουμε ως Επιτροπή για να ε, δώσουμε μια απάντηση στους αναφέροντες αφού έχουμε ακούσει και τις απόψεις των υπολείπων που θα ακολουθήσουν. Πάμε λοιπόν, προχωράμε πιο κάτω. 251 του 12 και 260 του 12. Την πρώτη θα την παρουσιάσει μία ένωση από το Λουξεμβούργο και η δεύτερη είναι από μία Πολωνέζα επίκο σχετικά πάλι με την κακομεταχείριση των ζώων. Τώρα, όσον αφορά την εκπροσώπηση αυτών των αναφορών, δεν υπάρχει κανείς από τους αναφέροντες. Ε, θα δώσω όμως το λόγο στην αρμόδια της Επιτροπής, την κυρία Μαργκερίτ Κούσμαν. Καλημέρα σας ε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας δώσω την απάντησή μου στα πολωνικά. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη ο έλεγχος σε ό,τι αφορά ε, τα κατοικίδια ε, ζώα, η μεταχείριση αδέσποτων σκυλιών και άλλα θέματα μπορεί να είναι ε, προβληματική κατάσταση. Έχουμε το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει την ανάγκη να γίνονται πλήρως σεβαστές οι απαιτήσει για την καλή υγεία των ζώων. Βέβαια, είναι δυνατόν να εφαρμόζονται διάφορες στρατηγικές επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, το άρθρο αυτό, παρότι υφίσταται, δεν αποτελεί νομική βάση. Τέλος πάντων, δεν ε, συνιστά απέτηση ε, για την κάλυψη όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την καλή μεταχείριση των ζώων. Άρα, δεν ρυθμίζεται το θέμα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Παραμένει λοιπόν αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει το έργο της ΒΕΒΕΦ που ζητά να εφαρμόζονται κάποια όροι για την προστασία και των αδέσποτων ζώων και τονίζει και τη σημασία της καταχώρησης ε, και της αναγνώρισης, ε, της επισήμανσης δηλαδή των ε, σκυλιών από τους κατόφτους Και το θέμα της εκτροφής είναι ένα ζήτημα. Έχουμε εγκρίνει κάποιους κανόνες το 2009, κάποιες αρχές. Αυτές ουσιαστικά αποτελούν πρότυπα που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όσοι καταρτίζουν νομοθεσία ε, ή αναλαμβάνουν να καταρτήσουν ε, κάποιας, κάποια μαθήματα επιμόρφωσης. Προβλέπονται επίσης κάποια ελάχιστα κριτήρια για την ε, φροντίδα που πρέπει να παρέχεται στα ζώα αυτά. Τα κράτη-μέλη όμως το καθένα από μόνο του και ως μέλη της βέβαια μπορούν να αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα, αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές στη δική τους επικράτεια και ανάλογα με τις ε, περιστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια συνεχίζει και θα συνεχίσει και στο μέλλον να συνεργάζεται με την Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων για το θέμα αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά νέες στρατηγικές, ε, στρατηγική για την ευζοία των ζώων από το 2012 έως το 2015. Θα εκπονήσει μια μελέτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ευζοία σκυλιών και γατιών που είναι αντικείμενο εμπορική δραστηριότητα. Όταν ε, δημοσιευθούν τα αποτελέσματα τη μελέτη, ε, η Κομισιόν ε, θα εξετάσει το ενδεχόμενο, εφόσον βέβαια αυτό χρειάζεται, του να προβεί σε περαιτέρω μέτρα. Βέβαια, πάντοτε λαμβάνοντα υπόψη την αρχή τη αναλογικότητα και την αρχή τη επικουρικότητα. Επίσης, ό,τι αφορά κάποιες προσδοκίες που μπορεί να έχει η κοινή γνώμη ή οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, θέλω να σας πω ότι περί τα τέλη Οκτωβρίου θα διοργανωθεί μια πρώτη ευρωπαϊκή ε, διάσκεψη για την ευζοία των ε, γατιών και των σκυλιών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα απορίσματα της μελέτης και τα αποτελέσματα αυτής της διάσκεψης η μελέτη θα είναι του χρόνου ε, έτοιμη πιστεύουμε, θα αποτελέσουν λοιπόν τη βάση για το δικό μας προβληματισμό για το θέμα αυτό στο μέλλον. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει και άλλες δράσεις για να υποστηρίξει την παροχή ε, τακτικών πληροφοριών ε, και την πρόθεση εκπαιδευτικών στρατηγικών για την καλή των ζώων. Μεταξύ άλλων, σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς όπως για την ε, δημιουργία ενός ε, δικτυακού τόπου που λέγεται Καρόντορ και είναι ένα ενημερωτικό ιστότοπος όπου γίνονται κάποιες προσπάθειες για να προωθηθεί η υπευθυνότητα ε, των ιδιοκτητών κατοικιδίων ζώων. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο να λάβει το λόγο για αυτές τις δύο αναφορές. Νομίζω ότι και εδώ, όπως σα είπα και προηγουμένως, ε, ισχύει το ίδιο εκ μέρου τη επιτροπή. Αυτά που μα είπε η κυρία Κούσμαν ήταν λεπτομερή, ήταν σωστά και δείχνουν και μία προσωπική εμπλοκή. Πιστεύω βέβαια ότι θα πρέπει να ε, δούμε και τι λέει το άρθρο 13, το οποίο προχωράει πολύ πιο πολύ από αυτά που κάνουμε. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να παρέμβει σε, ένα, σε τέτοιου είδου ε, περιστατικά. Ε, αυτά είναι θέματα εθνικής αρμοδιότητας. Όπως σας είπα λοιπόν και προηγουμένως, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ε, στις άλλες ε, δύο αναφορές και στο τέλος θα κάνουμε την αξιολόγησή μας και θα δούμε πώς θα καταλήξουμε. Επ' αυτού του θέμα για την 12.54 54 του 12 δίνω το λόγο την επόμενη αναφέρουσα είναι μια γαλίδα υπήκος ε, γαλλικής ηθαγένειας που αναφέρεται και αυτή πάντα ε, στο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ζώων. Παρόν όμως είναι ε, παρούσα η Μπέικ Μπάκμαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ζητούμε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία την προστασία των ζώων. Η εν νομοθεσία Ε, πρέπει να πούμε ότι είχε ως αποτέλεσμα να υιοθετηθούν διάφορα μέτρα θετικά και να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά κάποια από αυτά τα μέτρα ε, δεν είναι αποτελεσματικά γιατί δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Πρόσφατα άλλωστε αυτό το παραδέχτηκαν και οι Ευρωπουλευτέ. Η αναφορά μας λοιπόν ζητά βράχη πρόθεσμα τη δημιουργία μιας εξεταστικής επιτροπής ε, για την πραγματική κατάσταση των ζώων στην Ευρώπη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Επίσης, Ζητούμε να γίνει μια έρευνα σε ό,τι αφορά τις προκαταλήξεις ε, και τα τραύματα των Ευρωπαίων πολιτών, ε, τα ψυχικά τραύματα όταν βλέπουν ε, αυτά τα παραδείγματα κακομεταχείρισης, κακοποίησης των ζώων. Πρόκειται για ψυχικά τραύματα που ορισμένους πολίτες τους οδηγούν στο να ε, βγουν εκτός νόμου κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να απελευθερώνουν ε, κάποια πειραματόζωα από τα εργαστήρια κτλ. κτλ. Ζητούμε επίσης ε, να υπάρξει μια επιτροπή η οποία θα αναλάβει να ασχοληθεί με το σεβασμό της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των ζώων. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, μέσω πρόθεσμα ζητούμε να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για την κατάσταση και την προστασία των ζώων και ίσως ε, μακροπρόθεσμα τη δημιουργία αυτόνομων αποκλειστικών δομών για την ε, κατάσταση των ζώων και την προστασία των ζώων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Και όπως και τις προηγούμενες αναφορές ε, δεν είναι καθόλου προσαρμοσμένη και σωστή απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ μιλάμε για δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να δουν εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως μας μιλάει για το άρθρο 13, για την ευζοία των ζώων και συγκεκριμένα σκυλιών γατιών. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η κυρία Γκούσμαν, εκ μέρους της Επιτροπής. Sí, Madame la Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η απάντηση της Επιτροπής ε, είναι σχεδόν ταυτόσιμη με την προηγούμενη απάντηση που σας έδωσα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει νομική βάση για να ε, αναλάβει δράση. Πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα. Το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει τέλο πάντων ε, προβλέπει κάποιες απαιτήσει για την καλή μεταχείριση των ζώων. Άρα, και στα κράτη-μέλη, αυτά έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για να εφαρμόσουν τα σχετικά μέτρα. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αντιδράσει. Ευχαριστώ. Διόλου δεν συμφωνώ με αυτά που άκουσα, διότι το άρθρο 13 της συνθήκης της Λισαβόνας λέει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις της προστασίας των ζώων και όταν υποφέρει ένα ζώο πάει να πει ότι δεν ευημερεί, δεν ε, ε, προστατεύεται. Τα ζώα είναι ευαίσθητα όντα, άρα πρόκειται για κακή θέληση αν δεν θέλουν να... κακή πίστη δηλαδή αν δεν θέλουν να αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται. Εγώ ε, απευθύνω χαιρετισμό στην κυρία Όλτενμπουργκ που είναι ε, πρόεδρος του οργανισμού ε, για την προστασία των ζώων εδώ στην Ευρώπη κτλ. Και, και όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει αναφορά που συνυπογράφεται από 20.000 αναφερομένους στην Ισπανία. χιλιάδες λαγωνικά θανατώνονται από τους ε, ιδιοκτήτες τους όταν πια δεν ε, είναι ικανά να ε, κυνηγήσουν. Θα πρέπει να δείξουμε και εικόνες ίσως για να ευαισθητοποιηθούν επιτέλους και αυτή της Κομισιόν. Έχω δει εγώ και ταινίες και φωτογραφίες και είναι ανυπόφορες. Οι κυνηγοί διαθέτουν λαγωνικά για να κυνηγούν. Εντάξει, μπορεί να είναι κανείς αντίθεση με το κυνηγή. Τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν τα λαγωνικά αυτά δεν είναι πια αρκετά ικανά. Αισθάνονται οι ε, κυνηγοί οι ίδιοι ανίκανοι να κυνηγήσουν και τότε τα τιμωρούν. Τι πάει να πει αυτό? Είναι η τεχνική του πιάνου. Κρεμούν το λαγωνικό από ένα κλαδί με ένα σκηνή κοντό. Ίσα ίσα να μπορεί να κουμπάει τα πόδια του και το ζώο σιγά σιγά όταν χάνει τις δυνάμεις του απαγχωνίζεται ή τους κάνουν τα μάτια ή τα πετάνε ζωντανά μέσα σε πηγάδια και άλλα. Μπορώ να σας φέρω και εικόνες, μα συνεχίσω τις περιγραφές αυτές. Καλά, ωραία, η Κομισιόν λέει δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά κάποια στιγμή να σταματάμε μας λέει παραμύθια. Εγώ γνωρίζω ποιες είναι οι δυσκολίες που προκύπτουν από την κυριαρχία των χωρών μερών. Αν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέρει να επιβάλλει τους κλοβούς ορνήθων έτσι ώστε οι όρνηθες να μπορούν να μεταφέρονται με σε μεγαλύτερη γαλήνη κτλ. Πολύ καλά. Γιατί δεν μπορεί, μπορεί να αντιδράσει όταν σημειώνονται περιστατικά ε, ζωοκτονίας ή τέτοιες ε, σκηνές απίστευτης σκληρότητας και καμιά φορά μπροστά και στα παιδιά των κυνηγών. Γνωρίζω και άλλες χώρες όπου οι ε, κυνηγοί σέβονται τα ζώα τους. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η βάρβαρη μεταχείριση των λαγωνικών και των κυνηγετικών ε, σκύλων γενικά. Δεν έχει σχέση αυτό με το κυνήγι. Πρέπει να σταματήσει, να πάυσει αυτός ο βασανισμός των λαγωνικών. Όλοι μιλάνε γι' αυτό. Πρόκειται για εκατομμύρια λαγωνικά, για εκατομμύρια κυνηγετικά σκυλιά. Δεν κατανοούν οι άνθρωποι πλέον γιατί η Ευρώπη αφήνει ατιμόρυτες τέτοιες πράξεις. Ζητώ λοιπόν, απαιτώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ευνοϊκή συνέχεια στην αναφορά και να πάει να εξετάσει και επιτόπου αν χρειάζεται τι βάρβαρε αυτέ κοινέ μεταχείριση των ζώων. Και πολύ ευχαριστώ να μαζί σα. 20.000 υπογράφουν την αναφορά αυτή και έχουν το δικαίωμα να ακουστούν και ζητούν απάντηση. Μην κρυφτείτε πίσω από την αρμοδιότητα των χωρών μελών. Παρά είναι εύκολο αυτό. Μην αφήσετε τους κυνηγού να μας επιβάλλουν τα δικά τους, το δικό του νόμο. Δείξτε, δώστε μια αξιοπρεπή εικόνα της Ευρώπης και καθίστε να διαβάσετε σωστά το άρθρο 13 Τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Πολύ ωραία. Ε, δεν βλέπω να έχει δει κανεί άλλο το λόγο. Η συνάδελφο Χόκεν. Just a little point to the commission. Για την Κομισιόν. Σύμφωνα με αυτό το 13 που ακούστηκε τώρα κατά επανάληψη είναι εδώ το άρθρο, είναι αρμοδιότητα δική μας να κάνουμε κάτι. Ε, δεν εμπίπτει σε αυτό το «Α, δεν έχω αρμοδιότητα». Είναι μέσα στη συνθήκη, άρθρο 13. Δεν είναι εύκολη υπόθεση βέβαια, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αμελείται ε, ή παραμελείται αυτό το άρθρο 13. Κοιτάξτε, θέλω μόνο να επιβεβαιώσω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Δηλαδή το άρθρο 13 είναι απόλυτα σαφές. Η Επιτροπή δεν μπορεί να αρνηθεί ότι στη συνθήκη μας γίνεται λόγος για την καλή διαβίωση των ζώων και η μόνη αιτιολογία της Επιτροπής είναι ότι η ζωοτομία και η κτηνοβασία είναι μέρος της καλής διαβίωσης των ζώων. Πολύ ωραία. Να βγει κάτι τέτοιο στον τύπο και μάλιστα λίγο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Για να δούμε. Αναφέρθηκε το θέμα της κτηνοβασίας. Δεν ξέρω, έχετε δει ταινίε με αυτό το αντικείμενο που είναι ελεύθερο προσβάσιμο στο διαδίκτυο. Το ξέρετε αυτό. Εδώ μιλάμε για ευρωπαίους πολίτες που αντιμετωπίζουν ψυχικά τραύματα όταν δουν κάτι τέτοιο, ε, αυτή του είδους την κακοποίηση των ζώων. C'est tout à fait Είναι καθόλου η αρμόζουσα η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Asking to Mr. Law if we can go to, ask τον κύριο Λόου, αν ε, μπορούμε να ζητήσουμε μια γνώμη. Τέλος πρέπει να το σκεφτούμε. Μπορούμε να ζητήσουμε μια γνωμοδότηση. Λοιπόν, ε, μπορούμε νομίζω να περάσουμε στην τελευταία αναφορά και μετά να τις εξετάσω από κοινού όλες αυτές τις αναφορές. Κύριο Σάκταρ είναι εδώ. Madam Chair and honourable members, my name is Zaho Akhtar and on behalf of Animal Δήμαρχο άκτα λέγομαι από ε, την οργάνωση Animals Angel. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που μας δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Η πρόεδρος μας, κυρία Κρίστα Μπλάνκα, δεν μπορούσε να έρθει λόγω ασθενείας ε, σήμερα. Ε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οκτώ μήνες πέρασαν οπότε αρχίσαμε να συλλέγουμε υπογραφέ και έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο, εκατομμύριο 100.000 υπογραφέ από όλα τα κράτη για την αναφορά μα 971-2012. Ε, θέλουμε πραγματικά να αναλυφθεί δράση για να έχουμε οκτάωρο ε, περιορισμό ε, στο χρόνο ταξιδίου των ε, ζώων που μεταφέρονται προ σφαγή. Υπάρχουν ζώα που μεταφέρονται χωρίς επαρκή τροφή, νερό, με πάρα πολύ κακές συνθήκες. Έχουμε λάβει πάρα πολλές καταγγελίες και δείχνουμε και πάρα πολλά στοιχεία από την Animal Angels που το πιστοποιούν αυτό. Ε, προβλέπεται η μεταφορά ζώων από την Ευρωπαϊκή για πολλές μέρες. Ε, το θέμα δεν είναι μόνο όμως ότι δεν υπάρχουν σωστά νομοθεσία, Όσο ε, έχει αυτή τη στιγμή η νομοθεσία δεν είναι εφικτό να αποτρέψει τις καταχρήσεις, ακόμη δηλαδή και αν εφαρμοζόταν. Ένα εκατομμύριο λοιπόν, 103.248 συμπολίτες μας ζήτησαν αλλαγή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει αλλαγή, έχει υπογράψει την ε, γραπτή δήλωση πέρυσι το Μάρτιο. Περισσότεροι βουλευτές την υπέγραψαν αυτή τη δήλωση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης επίσης ζητά να υπάρξει αλλαγή. Ε, επίσης οι ε, κτηνίατροι στην Ευρώπη το ζητούν λυπούμαστε που η ομόφωνη φωνή των πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν λαμβάνεται υπόψη από την Κομισιόν. Μετά την γραπτή δήλωση την περσινή του Κοινοβουλίου, πάνω από 50 ερωτήσεις ε, κατατέθηκαν από ευρωβουλευτές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι απαντήσεις που έλαβαν νομίζω ότι δείχνουν στην καλύτερη περίπτωση αδιαφορία, απάθεια ή και έλλειψη κατανόησης για το αντικείμενο των ερωτήσεων. Εμείς λοιπόν ε, ζητούμε η Επιτροπή σας να επιληφθεί ε, με τον τρόπο με τον οποίο κρίνει βέλτιστο, να ζητήσει ε, ίσως ενημέρωση από την Κομισιόν, μέσω του Solvit, με οποιαδήποτε άλλη δράση μπορεί να αναλάβει για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να δοθεί απάντηση σε αυτή την αναφορά. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η μεγαλοσύνη των εθνών και η ηθική πρόοδος κρίνεται από το τρόπο που αντιμετωπίζονται τα ζώα. Αυτό είπε ο Γκάντι. Βλέπουμε όμως ότι παρά το ότι ε, υπάρχει ε, δυνατότητα, ε, υπάρχει αυτή η θετική δάδα που ε, κρατούν οι πολίτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν την έχει, δεν εισακούεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ εξ μέρους της Animals Angels. Thank you to you. The floor to... Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σίμωνιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω την γραπτή απάντηση της Κομισιόν, αλλά για την διάρκεια των μεταφορών των ζώων στην Ένωση υπάρχει εδώ και καιρό η σχετική νομοθεσία. Η, έχει υποβάλει, έχει εκκρίνει μάλλον έκθεση τον Νοέμβριο 2011 η Κομισιόν για τις μεταφορές ζώων γενικότερα και διάφορες επιστημονικές και κοινωνικο-οικονομικές πτυχές. Η θέση που παραμένει ίδια της Κομισιόν το 2011 είναι ότι δεν προτίθεται να προτείνει τροποποίηση στην νομοθεσία διότι θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμα από την υπάρχουσα νομοθεσία πολλά τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν και δεν σημαίνει ότι θα βελτιωθεί η προστασία των ζώων αν ψηφιστεί νέα νομοθεσία. Τώρα, για να συμπληρώσω τα όσα έχουμε υποβάλει εγγράφο, από το 2011 έχουμε ξεκινήσει συγκεκριμένες δράσεις που δεν θίγουν με την νομοθεσία, αλλά άπτονται άλλων μη νομοθετικών πτυχών. Απόφαση λοιπόν της Κομισιόν η οποία εγκρίθηκε για τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες μέλη προβαίνουν στους ελέγχους, τον τύπο των παραβάσεων που σημειώνουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι επιτρέπει στην Κομισιόν να κατανοήσει καλύτερα τι συμβαίνει από πλευράς δηλαδή προσπαθειών των χωρών μελών να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία για τις μεταφορές των ζώων. Επίσης, καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναπτύξουν ορθές πρακτικές για τη μεταφορά των ζώων. Υπάρχει και σχετικός οδηγός για τη μεταφορά των βοηδών που μάλιστα έχει ενημερωθεί, έχει επικαιροποιηθεί καθώς επίσης και για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μεταφορά των ζώων. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια τεχνική εργασία, συνεδριάσεις που συνέχονται τακτικά εμπειρογνωμόνων για την ε, συγκεκριμένη μελέτη των διαφόρων τομέων, τακτική επιθεώρηση το τι πράττουν οι χώρες μέλη για την εφαρμογή της νομοθεσίας και όπου αυτό απαιτείται κινούνται και διαδικασίες προσφυγής για παράβαση. Αυτά και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Άλλο παρακαλώ, επιτιμεί κάποιο άλλο το λόγο. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν συνάδελφοι που επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Ε, ο Ετών για να απαντήσει. Thank you for your response. And, um... Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ναι, μεν ε, ψηφίστηκε έκθεση το 2011. Πολλά έχουν γίνει από τότε, γιατί το θέμα είναι αρευστό. Πέρσι, στις 6 Ιουνίου 2012, κατατέθηκαν οι 1,1 εκατομμύριο υπογραφές, καθώς επίσης και μια γραπτή δήλωση από πέρσι, το 2011. Πολλά έγιναν λοιπόν από τότε, σε μια κίνηση προς τα εμπρός, Ο αξιότιμος επίτροπος λέει ότι υπάρχει θέμα υποβολής αναφορών από πλευράς χωρών μελών. Όμως σε απάντηση που δόθηκε από την Κομισιόν σε ερώτηση ευρωβουλευτών, η Κομισιόν είπε ότι δεν υπάρχει τρόπος να γίνουν γνωστά τα διαμυφθέντα. Στάθηκε επιστολή και όταν ρωτήθηκε εάν έγινε η ερώτηση, δηλαδή όταν, αν θα υπάρξει συνέχεια, δεν υπήρξε απάντηση. Δεύτερον, είπατε ότι υπάρχουν κατευθυντήρε γραμμές για ορθές πρακτικές. Αυτό όμως στην βάση της υποθέσεως ότι λειτουργεί η ισχύουσα νομοθεσία. Μπορεί μεν κανείς να προσπαθεί να βελτιώσει την εφαρμογή. Από την άλλη μεριά, οι έρευνες που κάνουν οι ομάδε μας σε όλη την Ευρώπη δείχνουν ξανά και ξανά ότι ακόμα και με τη σωστή επιβολή των ορθών πρακτικών, η νομοθεσία δεν αρκεί για να, για να ελαφρύνει τα βάσανα, τα βάσανα των ζώων. Υπάρχουν ζώα που μεταφέρονται για ημέρες ολόκληρες, επάπειρον σχεδόν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν λοιπόν άλλες ε, παρεμβάσεις από ό,τι βλέπω. Εσείς δεν είστε μέλος, εδώ η συζήτηση αφορά τα μέλη. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τις αναφορές τις οποίες εξετάσαμε και τα ερωτήματα που ετέθησαν, Νομίζω ότι όλα αυτά απορρίφθηκαν από την ε, Επιτροπή γιατί μας είπε ότι δεν είναι αρμόδια. Κυρίως όσον αφορά στις ε, αναφορές ε, που έχουν σχέση με, το μη επίκαιρο του όλου θέματος. Αλλά ξέρετε, πάνω από 1.300.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει αυτήν την αναφορά και αναφέρονται πέρα από όλα και στο θέμα της μεταφοράς των ζώων σε σχέση πάντα με την καλή διαβίωσή τους. Εκεί λοιπόν η Επιτροπή λέει ότι η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει να διασφαλίζει ε, κανείς την καλή διαβίωση των ζώων. Όσον αφορά όμως το θέμα το οποίο συζητάμε, ε, το θέμα της ε, κακομεταχείρισης και της βίας που ασκείται έναντι στα ζώα, ε, δηλαδή ε, την ε, ζωοτομία για επιστημονικούς λόγους. Γι' αυτό το θέμα η Επιτροπή λέει ότι δεν εμπίπτει στις δικές της αρμοδιότητες και λέει επίσης ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη αποφασίσει τροποποιώντας την προηγούμενη νομοθεσία με παρεμβάσεις ε, τα οποία έχουν αμβλύνει κατά κάποιον τρόπο τις ε, παρεμβάσεις έναντι των ζώων. Αλλά δεν αποκλείεται η ζωτομία τελείως για επιστημονικούς ε, σκοπούς. Και γι' αυτό το λόγο, όπως σας είπα, εμφανίστηκαν όλοι αυτοί οι πολίτες οι οποίοι υπέγραψαν αυτήν την αίτηση. Ένα άλλο θέμα αφορά στην κακομεταχείριση των ζώων, είτε είναι κατοικίδια ζώα, είτε είναι αδέσποτα ζώα είτε οποιασδήποτε άλλου μορφής. Σύμφωνα λοιπόν με την Επιτροπή και πάλι ε, δεν είναι αρμόδια γι' αυτά, δεν εμπίπτουν άμεσα στις ε, δικές της αρμοδιότητες. Αναφέρεται λοιπόν η Επιτροπή στο άρθρο 13 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο αποδίδει κάποιες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλή διαβίωση των ζώων, ε, κυρίως ε, για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν, όπως σας είπα, στην καλή διαβίωση των ζώων. Ε, στο θέμα της, του κυνηγιού, της μεταφοράς των ζώων. Αυτή είναι οι τομείς ε, όπου πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια έχουν εκχωρηθεί δηλαδή οι αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι αυτηρές καταγγελίες, δεν μπορούμε να μην προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Στο κάτω-κάτω αυτή είναι η δική μας ε, η δουλειά. Να προσπαθήσουμε να δώσουμε έτσι μια πιο ευρεία ερμηνεία, μια ερμηνεία που να αφορά κατά κύριο λόγο το άρθρο 13 που όπως σας είπα αναφέρεται στην καλή διαβίωση των ζώων. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να ζητήσουμε από την Αρμόδια Επιτροπή να ερμηνεύσει σωστά το άρθρο 13. Και επίσης μπορούμε να απευθυνθούμε και εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεσα με περώτηση στην Ολομέλεια. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά ε, δεν είναι ότι δεν έχει καμία πολύ αρμοδιότητα όπως θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει από αυτά που είπε σήμερα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το 2012 θέλησε να παραθέσει ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών όπου εκεί φαίνονται ποιες αρμοδιότητες ε, και ποια μέτρα μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλή διαβίωση των ζώων. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε μία μελέτη ε, δύο ετών. Επειδή λοιπόν τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μία αναφορά την οποία υπογράφουν τόσοι πολλοί πολίτες, πρέπει να ρωτήσουμε την Επιτροπή τι έχει κάνει σχετικά με αυτή τη μελέτη. Μήπως θα πρέπει λιγάκι να επιταχύνει και σε τελική ανάλυση ας μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε ορισμένες αξίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δηλαδή εδώ δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια ε, μπροστά σε τόσο ε, ιδεχθείς πράξεις όπως αυτές που αναφέρθηκαν. Η δική μου λοιπόν η πρόταση είναι η εξής. Να ζητήσω από εσάς τους συναδέλφους ε, να τοποθετηθείτε, να μας πείτε κατά πόσον συμφωνείτε με το να παρουσιάσουμε, να καταθέσουμε μια προφορική επερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το άρθρο 13, όπως επίσης και για τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει σχετικά με την προστασία των ζώων. Δεν βλέπω να υπάρχουν διαφωνίες. Άρα δηλαδή θεωρώ ότι εγκρίνεται αυτή την πρότασή μου και ευχαριστώ πολύ τους ε, ετούντες που μας παρουσίασαν αυτή την αίτηση και ευχαριστώ επίσης ε, το 1 εκατομμύριο περίπου 200.000 άτομα που απευθύνθηκαν σε εμά για να μας ε, επισημάνουν το θέμα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι η 1040 του 2012 από έναν Βρετανό πολίτη ε, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της συμβασής του Άρχους από τη Βρετανική κυβέρνηση. Και αυτή, ε, για αυτήν θα μας ενημερώσει η κυρία Τζέν Γκριν, ε, στην οποία δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να διαβάσουμε τη δήλωση. Διότι δεν μας επιτρέπεται να λάβουμε, ε, συμμετάσχουμε στις αποφάσεις για το περιβάλλον, για zero waste και για έργα υποδομής για την συλλογή των απορριμμάτων. Πολλές ε, δημοτικές αρχές προχωρούν με ιδιωτική με ιδιωτικό κεφάλαιο στη δημιουργία υποδομών για τη συλλογή των απορριμμάτων. Για να συμμετάσχει το κοινό στις ε, λήψεις αποφάσεων είναι μέσω του, people, του public planning process. Ωστόσο, η εμπιστευτικότητα, η μυστικότητα που ε, περιβάλλει τις ε, ενέργειες αυτές καθιστά δυσνόητο για το κοινό το τι γίνεται. Ενώ αυτοί έχουν στη διάθεσή τους δικηγόρους, το κοινό που επιθυμεί να αμφισβητήσει τις εξελίξεις αυτές δεν έχει τους πόρους για να προβάλλει τα επιχειρήματά του. Η κυβέρνηση του Ενωμένου Βασιλείου δέχθηκε ότι είναι απαραίτητο να δοθεί δικαστική, ε, δηλαδή νομική βοήθεια ε, στους ενδιαφερόμενους. Όμως η υπόθεση της μυστικότητας για τις λεπτομέρειες θα πρέπει να αρθεί και θα πρέπει να δοθεί νομική συνδρομή για αυτούς που ε, ενδιαφέρονται. Τις τελευταίες δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει δώσει σε, έχει σε πραγματική επανάσταση για την συλλογή των απορριμμάτων. Χωματερές κλπ. Για, το, για την ανακύκλωση, το composting κλπ. Και έτσι να κλείσει ο κύκλος στην οικονομία. Η ατζέντα ε, θα, θα εκπαιδευτεί και άλλο. Οι περισσότεροι πολίτες ενδιαφέρονται να υπάρξει ανακύκλωση και υπέρ του περιβάλλοντος και για να εξοικονομηθούν χρήματα. Φτάνουν ορισμένες κοινότητες και στο 70% της ανακύκλωσης με πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτές που δεν έχουν ανακύκλωση. Και βεβαίω επωφελούνται και από το εισόδημα που τους προσφέρει η ανακύκλωση. έτσι ώστε να υπάρχει ένα εύκαμπτο σύστημα. Βεβαίως, αυτές οι συμβάσεις PFI δεν ανταποκρίνονται στις αλλαγές που σημειώνονται στον κόσμο της ε, συλλογής των απορριμμάτων. Φτάνουν να κοστίζουν 49 εκατομμύρια ε, λίρες οι ε, απαρχαιωμένες αυτές συμβάσεις. Και τελικώς καθίσταται ακριβότερη η ανακύκλωση από το να απορρίπτονται στις ε, χωματερές. Το Ενωμένο Βασίλειο έχει επενδύσει σε μεγάλες εγκαταστάσεις καύσεως. Υπάρχει μάλιστα υπερχωρητικότητα στο Ενωμένο Βασίλειο. Δεν χρειάζεται να φτιαχτούν άλλα. Καλύτερα να αυξηθεί η ανακύκλωση. Προσφέρει πολλά ωφέλη. Τώρα, έτσι λοιπόν για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους, οι πολίτες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις επιλογές που κάνουν τα Δημοτικά Συμβούλια για τις μεθόδους ε, διαχείρισης των σκουπιδιών. Όμως δεν ακούγονται οι φωνές των πολιτών, διότι το λόμπι των εγκαταστάσεων καύσεων, καύσεως είναι πολύ ισχυρό. Και έχουν προωθήσει την ιδέα ότι η μοναδική ε, ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από τις χωματερές είναι αυτή, η καύση δηλαδή. Παρόλο που διαμαρτύρονται οι τοπικές κοινωνίες, δεν υπάρχει πρόσβαση σε ξεκάθαρες προφορίες και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να δείξουν οι διάφορες κοινότητες ότι υπάρχουν και άλλες συναρτητικές επιλογές. Με συμβάσεις με τις εγκαταστάσεις καύσεως της τάξης των 30 ετών και με κόστος ενός δισεκατομμυρίου καθεμιά δεν προχωρεί. Τώρα υπάρχουν και ε, εγγυήσεις που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών για να φτιαχτούν κι άλλα. Τα Δημοτικά Συμβούλια αναλαμβάνουν σημαντικούς εμπορικούς κινδύνους, οικονομικούς κινδύνους, που δεν θα μπορέσει να αντίξει ο, ο ιδιώτης εταίρος. Μεταξύ αυτών και τον κίνδυνο να υπάρξει υπερχωρητικότητα ανακύκλωσης και επομένως και μαζί μάλιστα και τον κίνδυνο λέει της αλλαγής στην ε, περιβαλλοντική νομοθεσία. Για παράδειγμα φορολογίες για ε, το διοξείδιο του άνθρακα ή για την διάθεση στα ε, απορρίμματα κτλ. Αυτά δεν τα γνωρίζουν ε, οι τοπικές κοινότητε. συχνά. Οι δε προκηρύξεις σε εκδηλώσεις δεν ε, περιλαμβάνουν και διαβούλευση με το κοινό για το πώς γίνεται η στάθμιση των διαφόρων παραγόντων. Συχνά περιλαμβάνουν ιδιαίτερα πράγματα για τις ε, τεχνολογίες που χρησιμοποιείται κτλ. Και χρειάζονται χρόνια για να φτάσουν να γίνουν γνωστές οι διάφορες συμβάσεις και όταν πια είναι πολύ αργά για να μπορέσει να τις ελέγξει το κοινό. Ακόμα και οι φτωχότερε τοπικές ε, κοινότητες δεν λαμβάνουν νομική σύνδρομη για να μπορέσουν να ε, συμμετάσχουν σε δημόσιες έρευνες και τα λοιπά σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων. Οι δε πολίτες δεν έχουν καν το δικαίωμα της ε, έφεσης. συχνά το κοινό έχει την εντύπωση ότι βρίσκεται σε αντιδικία αντί να συμβάλλει. Επίσης δεν υπάρχει και χρηματοδοτική δυνατότητα των μικρών κοινοτήτων ακόμα και εάν ε, συλλέξουν ε, ε, πόρους είναι πολύ περιορισμένοι οι πόροι αυτοί όταν έχουν απέναντί τους έμπειρους δικηγόρους και τεχνοκράτες οι οποίοι πληρώνονται εκατοντάδες χιλιάδες λίρες από τα Δημοτικά Συμβούλια με μυστικές συμβάσεις. Εγώ μαθαίνω ότι η Σύμβαση Άρχους εγγυάται σε κάθε έναν το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που διαθέτουν οι δημόσιες αρχές και υποτίθεται ότι πρέπει να διαδίδουν. Και αυτό πρέπει να αρχίζει από πρώιμο στάδιο για να μπορέσει να, γίνει, να γίνονται και σχετικές προσφυγές. Εγώ προτείνω το Ηνωμένο Βασίλειο να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του για να δώσει πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε σχέση με τη διαχείριση της υποδομής, ότι τα θέματα τα οποία αναφέρω σήμερα εδώ πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος και να γίνουν αλλαγές στους εθνικούς ε, κανόνες, συστήματα και διαδικασίες. Επίσης, πολλές γιγάντιες συμβάσεις ε, με τις εγκαταστάσεις καύσης προχωρούν τώρα στη λήξη τους. Ζητώ λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ζητήσει να επιβληθεί μορατόριουμ στα έργα αυτά όσο καιρό θα διεξάγονται οι σχετικές έρευνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Ευχαριστώ πολύ. Από τις πληροφορίες που λάβαμε είναι δύσκολο να εντοπίσουμε πού είναι αυτά τα έργα. δεν εξακολουθεί να μην είναι ξεκάθαρο ε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αποφάσεων και κατά πόσον εξετάζεται το IPPC αυτή τη στιγμή. Επίση, η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου εγγυάται τη δημόσια συμμετοχή στη δικασία λήψεω αποφάσεων σε σχέση με αποτεφρωτέ μέσω δράσεων που εφαρμόζουν τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το θέμα είναι αν λαμβάνεται, θα ληφθεί απόφαση στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη χρήση της γης. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες, στοχευμένες πληροφορίες, σε ποιο στάδιο είναι αυτό το έργο δηλαδή, για να δούμε και τα πραγματικά περιστατικά και την νομική κατάσταση. Αλλά με βάση τις ε, παρατηρήσεις ε, της αναφέρουσας δεν βλέπουμε να υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας για τη δημοσία συμμετοχή ό,τι αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση. Βασίλειο όταν δεν γίνεται δεκτή από αποκάλυψη κάποιων πληροφοριών, υπάρχει διαδικασία προσφυγής. Δεν είναι ξεκάθαρο από τις πληροφορίες που παίρνουμε από την αναφέρουσα κατά πόσον έγινε αυτή η προσφυγή και τι αποτέλεσμα είχε. Αν υπάρξει προσφυγή στον Επίτροπο ε, αν υπήρξε προσφυγή στον Επίτροπο Ενημέρωσης δεν γνωρίζουμε, ούτε ξέρουμε αν ασχολήθηκε το αρμόδιο δικαστήριο. Υπάρχει και μία πρόσφατη απόφαση, ε, μάλλον τα πορίσματα του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C279-2012 που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη οι φορείς ε, που εκτός από τη διαχείριση κάνουν και άλλες, ε, αναλαμβάνουν και άλλες δράσεις, δεν υποχρεούνται να δώσουν πληροφορίες όπως λαμβάνουν σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες. Άρα να ληφθεί αυτό υπόψη. σε ό,τι αφορά πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά στήματα ενημερώθηκε η Επιτροπή για την υπόθεση C530 του 2011 για ε, το Ηνωμένο Βασίλειο. Γενικό Αγγελέα έχει προβεί σε κάποια συμπεράσματα τα οποία είναι χρήσιμο να ληφθούν υπόψη. Βελτιώσεις στο σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου έγιναν Δεν ξέρουμε αν θα ακολουθηθεί από το δικαστήριο η άποψη του Γενικού Εισαγγελέα. Αν ναι, θα πρέπει, επειδή είναι απαγορευτικό το κόστο σε ε, Ηνωμένο Βασίλειο, να ληφθούν μέτρα για τον ε, περιορισμό του κόστου. Νομική βάση πάντω δεν υπάρχει για να δημιουργηθεί ένα ειδικό σύστημα σαν αυτό που ζητά η αναφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ. να δώσω το λόγο στην κυρία Άουκεν και έχουν στήσει και άλλοι δύο συνάδελφοι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εδώ πρόκειται για δύο πράγματα. Το ένα είναι ένα γενικότερο ε, φύσεως ε, ερώτημα αφορά στους αποτεφρωτήρες. Ούτε στη Μεγάλη Βρετανία, ούτε στη Γερμανία υπάρχει ταύτιση των νομοθεσιών. Δεν είναι ίδιες οι νομοθεσίες ε, στις χώρες αυτές. Και στη δική μου τη χώρα μιλάμε για ορδές πυρομανών και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε κυρίως να γίνει είναι να υπάρχει ανακύκλωση και με βάση την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό που ενδιαφέρει βέβαια είναι η συμφωνία και η τήρηση της συνθήκης του Άρχους. Ο πολίτης με βάση τη συνθήκη αυτή έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται και αν το κρίνει απαραίτητο να ε, καταθέσει και μήνυση έναντι των κρατών. Πρέπει λοιπόν να παραμείνει αυτή η δυνατότητα ε, προσφυγής ε, στα δικαστήρια ακόμα και εάν δεν υπάρχει η πρόσβαση ε, σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει το θέμα να το αφήσουμε να τρέχει και από το πρίσμα των αποβλήτων και από το πρίσμα της ε, παραβίας της συνθήκης στο μέλλον θα πρέπει οι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε, τόσο σημαντικά θέματα όπως είναι το περιβάλλον. Και είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη απλά θέλουν να ξεφορτωθούν τους ε, πολίτες δίνοντάς τους λίγες πληροφορίες. Αυτή είναι μια καταπληκτική ε, αναφορά. Ευχαριστούμε την αναφέρουσα που ήρθε. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να μετακινηθεί και η Κομισιόν σε διάφορα επίπεδα. Καλησπέρα. Έρχομαι από την Κυπούσκοα, από την χώρα των Βάσκων, όπου δεν είναι μόνο τεχνικό θέμα διαχείριση των αστικών ελλημάτων και αποβλήτων, αλλά και ένα πολιτικό θέμα και έχει προκαλέσει και έντονη κοινωνική συζήτηση και τα περιβαλλοντικά ε, κοινοβούλια έχουν κατηγορήσει και καταγγείλει τις τοπικές αρχές. Αυτό το οποίο έχουμε μάθει όλη αυτή τη διαδικασία και είμαι και σύμβουλος σε ένα ε, δήμο, η ε, κυβέρνησή μας πρέπει να λάβει σε κάποιους μήνες κάποιες αποφάσεις για το σύστημα διαχείρισης αστικών λιμάτων, αποβλήτων που είναι αρμοδέτα των Δήμων. Αν λοιπόν κάτι μάθαμε με όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν κρατήσει μήνες και χρόνια είναι ότι η διαφάνεια σε ό,τι αφορά την μέρος των πολιτών ε, η δυνατότητα να ενημερώνονται και να συμμετέχουν οι πολίτες ε, στις διαδικασίες ε, είναι ένα θέμα το οποίο εφιστά την προσοχή της κοινή γνώμης σε αυτό το θέμα και γι' αυτό προσέχει πολύ περισσότερο το θέμα και η κοινή γνώμη αλλά και η Δήμη. Γιατί σε Δήμους που υπήρξε προσπάθεια να γίνουν ε, τα πράγματα έτσι στο πόδι γρήγορα, χωρίς συμμετοχή των πολιτών, χωρίς συζήτηση, δημιουργήθηκε κοινωνική αντιπαράθεση. Βλέποντας και ακούγοντας ε, αυτό που είπε αναφέρουσε και χαίρομαι που θέτει το ζήτημα αυτό, πιστεύω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διδαχθεί κάτι και θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί ώστε τα κράτη ε, σε ό,τι έχει να κάνει με την περιβαλλοντική διαχείριση και εδώ με τα αστικά λίματα και τα στερεά απόβλητα θα πρέπει να φροντίσει να υπάρξει μέγιστη δυνατή διαφάνεια καθώς και συμμετοχή των πολιτών και φυσικά και των δημοτικών αρχών στη λήψη αποφάσεων. Και νομίζω ότι στο θέμα αυτό υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη Βρετανία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να πω το εξή όσον αφορά αυτή την περίπτωση. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί η κατάσταση αυτή προκύπτει στη δική μου την εκλογική περιφέρεια, στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο αναφέρον προέρχεται από τα West Midlands. Αλλά είμαι και εισηγητή του Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι όλα αυτά πρέπει να είναι συμβατά με τη σύμβαση αρχού και γι' αυτόν τον λόγο ενδιαφέρομαι επίση ιδιαίτερα για την αναφορά αυτή. Νομίζω ότι ο αναφέρον καταθέτει μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, σωστά τεκμηριωμένη και παρακαλώ την Επιτροπή Αναφορών να την κρατήσει αυτή την αναφορά, να μην την κλείσει. Το θέμα είναι ότι το, ε, η υπόθεση έχει παραπεμπτεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα για να υπονομεύσουμε την ε, δικαστική διαδικασία που τρέχει. Το άλλο είναι το εξής. Από ό,τι φαίνεται, εκτός βέβαια αν ε, πει κάτι διαφορετικό ο αναφέρον, αν ε, δεν είναι κανείς πλούσιος ή αν δεν έχει πρόσβαση σε μυστικές πληροφορίες, οι δυνατότητές του για ε, να συμμετέχει δημοκρατικά σε διαδικασίες που τον αφορούν, αυτό είναι αδύνατο, παραδείγματο χάρη. Εάν θέλει κανείς να αμφισβητήσει μία απόφαση για μία μονάδα καύσης αποβλήτων ε, και δεν έχει κανείς ε, πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες που οδήγησαν στο να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, στο να η μονάδα, τότε πώς μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το όλο θέμα. Ε, χρειάζονται χρόνια, όπως λέει και ο αναφέρον, για να αποκτήσει κανείς ε, πληροφορίες που είναι απαραίτητες όμως για να ε, μπορεί κανείς να προχωρήσει. Αυτά υποτίθεται είναι εμπορικού συμφέροντος. Όμως αν υπάρχουν άνθρωποι σε τοπικό επίπεδο που για καθαρά δημοκρατικούς λόγους θέλουν να έχουν άποψη, να προγραμματίζουν τις αποφάσεις και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ε, μέσα από τα τοπικά συμβουλία. Τότε τι γίνεται. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για να παραμείνει ενισχύει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Για μένα αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι τους ανθρώπους αρνούνται την πρόσβαση σε πληροφορίες που αν τους τις έδιναν θα είχαν τη δυνατότητα να αμφισβητούν αποφάσεις που λαμβάνονται από τοπικά συμβούλια κυρίως για θέματα περιβάλλοντος. Και αυτά δεν περιορίζονται μόνο σε μικρές ε, κοινότητες. Τώρα όσον αφορά την νομική αρρωγή ε, ξέρω ο, ξέρω ποια είναι η απάντηση της Επιτροπής, όμως ε, παρόλα αυτά αυτό που ε, θα ήθελα λιγάκι να μας εξηγήσει η Επιτροπή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βλέπει να υπάρχει καμία παραβίαση από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου ε, όσον αφορά τους κανόνες συμμετοχής που αναφέρονται στην οδηγία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτό το περιθώριο της ε, διακριτικής ευχέρειας είναι προς όφελος εκείνων που κατασκευάζουν τον αποτεφρωτών, ενώ θα έπρεπε να είναι προς όφελος των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλω. Α, ναι, κύριε Ποστινάρου, με συγχωρείτε, σας ξέχασα. Ε, εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αναφορά και να πω κάτι που είναι προφανές. Στην επόμενη συνάντησή μας στο Στρασβούργο, στη Σύνοδο μάλλον, το Στρασβούργο, το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει σημαντικό νομοθέτημα που περιλαμβάνει τις αλλαγές στην οδηγία για τις μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου. Ο τρόπος με τον οποίο μέσω των τροπολογιών φαίνεται ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να ενισχύσει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της διαφάνειας για τις αρχές, να παρέχουν δηλαδή και στοιχεία για το ρόλο των πολιτών σε όλη τη διαδικασία. Να προσφέρουν και εναλλακτικέ τεχνικές λύσεις. Επίσης, πώς το Κοινοβούλιο απεφάσισε να περιγράψει και να καταγράψει την ανεξαρτησία του φορέα που μελετά την περιβαλλοντική, ε, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, επίσης την σύγκρουση συμφερόντων. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Επιτροπή Αναφορών που εγώ χαιρετίζω διότι φάνηκε πολύ ευχή όταν κατέθεσε τόσες πολλές σημαντικές τροπολογίες για την σχετική έκθεση και εγώ είμαι πεισμένος ότι όταν θα εγκριθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου στο Στρασβούργο οι χώρες μέλη μας και οι δημόσιες αρχές μας επιτέλους θα υποχρεωθούν να δρουν ορθά λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των πολιτών και όχι μόνο των επιχειρήσεων. Ελπίζω δε ότι η Κομισιόν επιτέλους θα εγκαταλείψει αυτή την ε, άτολμη τακτική της απέναντι σε όλες τις υποθέσεις που τίθεται υπόψη της Επιτροπής Αναφορών μας, αλλά και πραγματικά προσβάλλουν όλους όσοι πιστεύουν στην συμμετοχή των πολιτών, στην, μια προσπάθεια προστασίας των ε, ε, κοινοτήτων τους και επιλογής ε, περιβαλλοντικών λύσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που είπε ο κύριος Κάσμαν. Κοιτάξτε, εγώ συμμετέχω στο Worcestershire, στο Brace, σε αυτό το συγκεκριμένο project και δεν είναι μόνο το οικονομικό όπου δεν παίρνουμε απαντήσεις. Εγώ προσπάθησα να βρω κάποια στοιχεία, αλλά μάταια, διότι φαίνεται ότι όλα αυτά είναι μυστικά και η σύμβαση και όλα. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι σημαντικά. Ε, αυτός ο αποτεφρωτήρας ε, έχει κατασκευαστεί πάνω σε ένα χώρο από αποβλήτων που δεν είναι ακίνδυνος και διαρωτώ με πώς μπορεί να γίνει αυτό. Είναι ασφαλές. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στον χώρο αυτό υπάρχει ένα προστατευόμενο είδος και αντί να έρθουν σε επαφή μαζί μου, ξέρετε τι κάνανε. Έστειλαν ανθρώπους να πιάσουν αυτά τα πουλιά, το προστατευόμενο είδος, να τα βάλουν σε κλουβιά και το έκαναν αυτό παράνομα. Διότι για να το κάνει κανείς ε, κανονικά ε, θα έπρεπε να έχει άδεια. Ε, και αυτοί το έκαναν μυστικά. Έτσι λοιπόν κατά την άποψή μου Όλα αυτά ε, γίνονται συγκαλυμμένα και έχει έρθει πια η στιγμή να κατανοήσουν όλοι τι κάνει αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση επιτόπου. Nobody else? So I can go back to the petition. Mrs. Green for a reply. Yeah, I've been very ε, πολύ με ευχαρίστησε η όλη συζήτηση. Θέλω απλά να πω ότι έγινε κάποια αναφορά σε επιτρόπους ενημέρωσης, information commissioners. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν ε, την εμπορική επιστευτικότητα, τον εμπορικό απόρριτο να το ε, ξεπεράσουν αυτοί οι επίτροποι για η συγκεκριμένη περιοχή, το Χάλτμπρι, υπόθηκε εκεί ότι θα ληφθεί απόφαση 4 Οκτωβρίου, ας πούμε. Ε, και μπορεί για 5 χρόνια τώρα να... 15 χρόνια, μα θα έλεγα εγώ, έχει ξεκινήσει αυτό το θέμα. Καμία σύμβαση, καμία πιωματική υπόθεση δεν έχει δημοσιοποιηθεί, άρα δεν υπάρχει κανένα ε, συγκριτικό σημείο αναφοράς για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Πάντως σας ευχαριστώ, ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επισημάνατε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ και τους συναντέλφους για τη συζήτηση ε, που τα μισά τα άκουσα, τα άλλα μου τα είπανε ε, υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, άρα δηλαδή αυτή η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και να ξανασυζητηθεί, ε, προφανώς και μετά την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ας αφήσουμε λοιπόν ανοιχτή αυτή την αναφορά, περιμένοντας ε, να μας δοθούν περισσότερες πληροφορίες και σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης ε, στο δικαστήριο. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, συμφωνώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, διότι οφείλει να ολοκληρωθεί και η δικαστική ε, υπόθεση, αυτή, η υπόθεση ενώπιον του δικαστήριου. Εξάλλου, η νομοθεσία για την ε, πρόσβαση του κοινού στα επίσημα έγγραφα δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ε, ε, σύμβασης του άρχους και πρέπει να συμμορφωθεί. Έτσι λοιπόν υπάρχουν δύο λόγοι για να περαμείνει ανοιχτή η αναφορά. Μάλιστα. Συμφωνώ και εγώ, άρα κλείσει η συζήτηση για το θέμα αυτό και να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τη συνάδελφο που μας επισήμανε το θέμα και πάμε στο επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την έκθεση σχετικά με την διερευνητική επίσκεψη στη Δανία. Και εδώ ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, στη συνάδελφο Βέρτμαν. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Έχετε διαβάσει φαντάζομαι την έκθεση και θα ήθελα ε, να ξεκινήσω με ένα σχόλιο που αφορά αυτή τη συνάντηση. Είχαν προσκληθεί ο υπουργό ε, και ε, ο Γενικός Διευθυντής Αστυνομίας ή η, υπουργό, αυτή η καινούρια υπουργό ε, Εσωτερικών απάντησε και είπε ότι δυστυχώ δεν μπορούσε να έρθει ε, και πρέπει να την ευχαριστήσουμε που απάντησε. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με μια τεχνική εξήγηση. Υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά θέματα, ερωτήσεις που ετέθησαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Να δούμε λιγάκι ποιος είναι ο ρόλος μας ως Επιτροπή Αναφορών. πρέπει καλούμεθα να εξετάζουμε αυτά που μας λένε οι πολίτες, ενδεχόμενες παραβιάσεις της συνθήκης, ε, να απευθυνόμεθα σε όλες τις αρμόδιες αρχές, εθνικές, περιφερειακές, τοπικές. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ένας Ευρωπαίος πολίτης ε, μπορεί να καταθέσει μία αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις παραλάβουμε την αναφορά, αυτή την εξετάζει η Επιτροπή και η Επιτροπή την κρίνει παραδεκτή ή όχι. Τώρα, ε, τι είναι οι αποστολές επιτόπου. Οι αποστολές αυτές γίνονται με την έγκριση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι δηλαδή μια επίσημη αντιπροσωπεία η οποία αποτελείται από μέλη της Επιτροπής Αναφορών και αυτά τα μέλη της Επιτροπής ορίζουν και έναν επικεφαλής. Κατά κανόνα πρέπει να πω, διότι αυτό δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση, ε, Κατά κανόνα υπάρχουν και άλλα ε, μέλη ε, εξοφίτσιο ε, που προσπαθούν και αυτά να δουν αυτά που δεν γνωρίζουμε. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό για τους αναφέροντες να κατανοήσουν ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε μόνο με βάση πληροφορίες που μας έχουν δοθεί για θέματα τα οποία είναι σημαντικά. Και ε, εμείς δεν είμαστε δικαστές, ούτε και η Επιτροπή είναι δικαστήριο. Αυτό πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να αναφέρω ότι μας πλησίασε ε, η άλλη πλευρά, ένας από τους διάδικους αν θέλετε, ένας από, τους, από την άλλη πλευρά α, και όχι από τους αναφέροντες. Εμείς όμως συνήθως έχουμε να κάνουμε με τους αναφέροντες. Ας δούμε λοιπόν λιγάκι ε, ποιος είναι ο ρόλος μας. Μπορούμε να επισημάνουμε στις αρμόδιες αρχές ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα του οποίου πρέπει να επιληφθούν. Και αυτό είναι απόλυτα σαφές. Και πότε μπορούμε να το κάνουμε κυρίως ε, όταν παραβιάζεται η ενωσιακή νομοθεσία και αυτό αφορά βεβαίως και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσον αφορά λοιπόν την αντιπροσωπεία μας, ε, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία αλλαγή. Οι συνάδελφοί μου και εγώ συμφωνήσαμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω κυρία Πρόεδρε ότι προσβλέπουμε στη συνεργασία και στην ε, ε, βελτίωση της κατάστασης. Και έτσι φτάνω ε, στην κατάσταση που υπάρχει. Έχουμε λάβει αναφορές και οι αναφορές αυτές συζητήθηκαν το Φεβρουάριο και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας καταλάβαμε ότι είναι ιδιαίτερος επίγον να πάμε στην Δανία διότι θεωρούμε ότι η αναφορά αυτά, αυτή δεν αφορά μόνο τους αναφέροντες, ε, τους γονείς, ε, δανούς και μη δανούς. Ε, αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι τα παιδιά και η παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών. Αυτό τα πήραμε πολύ σοβαρά και αποφασίσαμε να πούμε σε επιτόπια έρευνα. Οι αναφέροντες ε, αναφέρουν ε, θέματα ε, που κατά δική μας άποψη πράγματι υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εδώ εντάσσεται και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως και η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Παιδιών και η Οικουμενική Διακήρυξη για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών. Θέλω λιγάκι να σας παρουσιάσω τη δομή αυτής της αποστολής Προσκαλέσαμε βέβαια και τον αρμόδιο Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης και τον επικεφαλής, ε, των διοικητή της αστυνομίας. Είχαμε ε, αποφασίσει να συναντηθούμε νωρίτερα για να έρθουμε σε επαφή με αυτούς. Βέβαια, ε, κανείς δεν ήρθε τελικά και είπανε αυτό λόγω των θερινών διακοπών. Εμείς είπαμε ότι είναι η πρώτη φορά όπου οι υπουργοί αρνούνται μία συνάντηση με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θέλω να σας πω ότι λίγες μόνο ημέρες μετά την αποστολή αυτή πήρα ένα σημείωμα ότι ο Υπουργός, η Υπουργός ε, Κοινωνικών Υποθέσεων προτιμήσε να παραμείνει στο σπίτι της, στον κήπο της και στην αυλή της. Και μετά από λίγες μέρες όμως βρήκε καιρό να δεχθεί την αντιπροσωπεία των Κινέζων. Κάτι δεν πάει καλά λοιπόν. Αυτή προτίμησε να παραμείνει όπως σας είπα στην αυλή του σπιτιού της. Και δυστυχώς και η νέα ή ο νέος υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων δεν κάνει και αυτός τίποτα, όπως ε, συνέβη από την αρχή και με την Υπουργό Εσωτερικών. Και αυτό θα το ψάξουμε. Όσον αφορά την κυρία Χέκερουπ, την Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων, ήδη από το 2007 το γνώριζε αυτό το πρόβλημα και πιστεύουμε ότι και ο Υπουργός Δικαιοσύνης γνωρίζει, ήδη το γνώριζε τότε το πρόβλημα. Δυστυχώς όμως ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν τοποθετείται από αυτού. Όπως είπαμε ήδη τον Ιούλιο, στη συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο. Εκεί συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη από το γραφείο του Υπουργού και τέθησαν αρκετές ερωτήσεις. Βεβαίως, αυτοί που ήταν παρόντες προσπάθησαν να απαντήσουν όσο καλύτερα μπορούσαν, αλλά όλοι μας συμφωνήσαμε ότι θα προτιμούσαμε να μιλήσουμε με τον Υπουργό. Γιατί σε τελική ανάλυση φύγαμε χωρίς να έχουν απαντηθεί πολλές μας ε, ερωτήσεις. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά δεν μπορούσαν να δώσουν καλύτερες απαντήσεις, δεν ήταν υπουργό, είναι στελέχη για συγκεκριμένους ε, τομείς. Και έτσι φτάνω σε αυτό που λένε οι αναφέροντες και να πω για άλλη μια φορά ότι στην έκθεσή μας, κυρία Πρόεδρε, αναφέρουμε μόνο τα πιο σημαντικά γεγονότα. Τα προβλήματα που εντοπίζουμε, όλα αυτά τα αναφέρουμε συνοπτικά. Είχαμε μια συνάντηση με τους αναφέροντες για πάνω από τέσσερις ώρες και είμαι σίγουρη ότι ο Κάρλος τα θυμάται αυτά. Εμείς δεν τολμήσαμε να πούμε τίποτα. Ήταν ιστορίες που ακούσαμε πραγματικά ανατριχιαστικές. Είχαμε το 90% γονιών μητέρων από τη Δανία, το 10% δεν ήταν Δανέζες και είχαμε και μερικούς μη Δανούς πατέρες. Εμείς από την αρχή καταλάβαμε ότι το πρόβλημα είναι βασικά η γονική ευθύνη που εισήχθη το 2007 Κατά την άποψή μας είναι σωστός αυτός ο νόμος, γιατί διασφαλίζει το παιδί να έχει επαφή και με, τα δύο, και με δύο γονείς και τούμπαλιν. Όσον αφορά όμως την πρακτική εφαρμογή, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που έχουν σχέση με την γονική μέρημνα. Όπως σας είπα προηγουμένως, ε, οι μητέρες δεν ήταν μόνο Δανέζες, ήταν και αλλοδαπές. Και υπήρχε και μια μικρή ομάδα αλλοδαπών πατέρων. Επιτρέψτε μου τώρα να μπω λιγάκι σε Αν μια μητέρα επιθυμεί να προστατεύσει το παιδί της από έναν βίαιο πατέρα, στο δικαστήριο δεν κρίνεται ο πατέρας, αλλά η μητέρα εκείνη κρίνεται γιατί υποτίθεται αυτή δεν συνεργάζεται κάτω από το πρίσμα του νόμου περιγονικής μέρης Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Αν κάποιος δεν μπορεί να προστατεύσει το παιδί του που είναι αντικείμενο βίας και μην ξεχνάτε τι ακούσαμε. Ένας, ε, ένας τέλεχος είπε ότι Μερικές φορές είναι καλύτερο το παιδί να πηγαίνει ακόμα και με έναν δύο ε, πατέρα. Και τίθεται το εξή ερώτημα. Ίσως επειδή είναι άνδρας ή μη, ίσως είναι επειδή είναι δανός. Ακόμα και δανείς συνάδελφοι είπαν ότι εδώ πρόκειται περί διακριτικής μεταχείρισης. Και θέλω να σας ε, πω ε, όταν έγινε η ερώτηση κατά πόσον υπάρχει διακριτική μεταχείριση η απάντηση είναι ότι δεν έχει καταγραφεί τέτοιου είδους διάκριση. Αυτά μας τα είπε ένας συνεργάτης ε, του ε, Ombudsman, του διαμεσολαβητή. Και κάτι άλλο πέρα από αυτό το θέμα με τον πατέρα. Πολλές αποφάσεις λαμβάνονται απλά επειδή έτσι συνηθίζεται. Δηλαδή, οι άντρες ε, δεν κρίνονται γιατί αυτό δεν συνηθίζεται, όμως από ό,τι φαίνεται συνηθίζεται να κρίνονται οι μητέρες που επιθυμούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Σε ορισμένες ε, περιπτώσεις, ε, με βάση το, την παράγραφο 215, οι γυναίκες φυλακίζονται με την κατηγορία της απαγωγής παιδιού. Τώρα, το θέμα του αν υποφέρουν τα παιδιά αυτό δεν πρέπει καν να συζητιέται διότι όπως είπα προηγουμένως είτε θα παραμείνουν με τον βίο πατέρα είτε ε, θα πάνε σε ένα είδο οικοτροφίου και μερικά από αυτά ε, δεν έχουν καθόλου πια την ευκαιρία να δουν τη μητέρα τους ε, ούτε και ε, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ούτε και αργότερα μερικές φορές μας είπαν μάλιστα ποτέ και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε σε άλλες περιπτώσεις, όπου η μητέρα θέλει να μετακινηθεί σε άλλη πόλη, χάνει την γονική μέρημνα απλά και μόνο, διότι πρέπει και ο πατέρας να έχει ε, επαφή με το παιδί. Και πραγματικά θεωρούμε ότι της απαγορεύεται να μετακινείται μόνο και μόνο λόγω αυτού. Γιατί δεν έρχεται ο πατέρας σε ε, μία πόλη πιο κοντά στο παιδί. Επίσης, η παράγραφος 35 του νόμου περί ε, κοινής γορικής ε, μέρημνας αναφέρει ο νόμος ότι αν το παιδί το επιθυμεί ε, μπορεί να καταθέσει στο δικαστήριο. Ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου τα παιδιά κατέθεσαν αλλά δεν άλλαξε τίποτα. Ο πατέρας εκλήθη να ακούσει την κατάθεση του παιδιού και η απάντηση που έδωσε στις περιπτώσεις αυτές ήταν ότι το παιδί λέει ψέματα, είναι υπό την πίεση της μητέρας και όλα πάνε μια χαρά. Και το ε, είπε τώρα ο πατέρας ότι το παιδί εξακολουθεί να θέλει να τον βλέπει και στις περισσότερες περιπτώσεις ο πατέρας πήρε και την αποκλειστική γονική μέρημνα. Σε άλλες περιπτώσεις το παιδί δεν ήθελε με τίποτα να επιστρέψει στον πατέρα μετά την ε, κατάθεση στο δικαστήριο σαφής παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού. Το κατάλαβε αυτό το παιδί και γι' αυτό πολλές φορές τα παιδιά αυτά ε, έφυγαν τρέχοντας. Και μετά υπάρχει και μια ομάδα παιδιών που πήγανε πίσω στη Δανία, κατ' ουσίαν όμως αυτό είναι απαγωγή. Και η κατάσταση είναι η εξή. Οι μητέρε φεύγουν από τη χώρα, σεβόμενε το νόμο. Ε, τα παιδιά καταγράφονται στα επίσημα μητρό ότι έχουν φύγει από τη Δανία. Οι μητέρε έχουν την αποκλειστική γονική μέρημνα και μετά οι δανικές αρχές αναδρομικά χορηγούν την κυδαιμονία στον πατέρα και με τον τρόπο αυτό ανοίγουν ουσιαστικά δίνουν το πράσινο φως για παγωγή. Σε μία περίπτωση ακόμα και ένας ε, διακεκριμένος νομικός αποφάντηκε ότι το παιδί δεν έπρεπε να, μάλλον ο πατέρας δεν έπρεπε να πάρει αναδρομικά την ε, μέρημνα ε, και ότι η μητέρα είχε φύγει νόμιμα από τη χώρα. Μετά υπάρχει και άλλη μια μικρή ομάδα μητέρων που παίρνουν ε, φάρμακα αναγκαστικά. Πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Για να καταλάβετε λίγο περισσότερο, ε, θα αναφέρω και κάποια συμπεράσματα. Έκανα μόνο αναφορά στα βασικά σημεία. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι δυσανάλογα βαρύ ο αντίκτυπο τη νομοθεσία τη Δανία για την μέρα των παιδιών. Οι Δανείοι πολίτε ε, και συγκεκριμένα οι άντρε πιο πολύ έχουν ε, το πάνω χέρι, ιδίω απέναντι σε μη Δανού επικόου που νιώθουν από τις ε, δανεικές αρχές να ε, υφίστανται διακριτική μεταχείριση. Θέλω να σας υπενθυμίσω κάτι το οποίο είπε ένας εκπρόσωπος του Δανού, συνηγόρου του πολίτη. Δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση, δεν έχει καταγραφεί ε, με τον τρόπο αυτό. Και μάλιστα τα δικαιώματα του παιδιού πολλές φορές δεν γίνονται σεβαστά, κάτι το οποίο διαπιστώσαμε. Οι μητέρες έχουν ε, την αίσθηση ότι η τρέχουσα δανεική νομοθεσία δεν ε, τους παρέχει ε, τη δυνατότητα να προστατεύσουν τα παιδιά τους από μια κακή συμπεριφορά από τον πατέρα. ακούσαμε διάφορες περιπτώσεις, οι μητέρες μόνο, δανές και μη ήταν αυτές οι οποίες απειλήθηκαν ή με την παράγραφο 250. Επίσης θέλω να σας πω ότι μας ενημέρωσαν για περιπτώσεις με έντονο ποινικό χαρακτήρα. Τις ε, παραδώσαμε στην εισαγγελία. Ε, θέλω να σας πω ότι έχετε και μία σειρά από συστάσεις, ε, τις οποίες εμείς έχουμε καταρτήσει. Θα ήθελα να σας πω δύο σημαντικά Πρώτον, ζητούμε η Δανία να ακολουθεί, να τηρεί τα ψηφίσματά της, ε, τις αποφάσεις που λαμβάνει και να εφαρμόσει την σύμβαση της ΧΑΙΣ για τις αστικές πτυχές ε, περί ε, διεθνούς αρπαγής παιδιών και επίσης να εφαρμόσει και την σύμβαση για την προστασία των παιδιών. Δεύτερον, θέλουμε να τονίσουμε ότι καλούμε επίσης μεταξύ άλλων να γίνει επίγουσα αναθεώρηση ε, και επανεξέταση των υποθέσεων επιμέλειας ε, και των ε, περιπτώσεων διεθνής αρπαγής παιδιών, ώστε να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και επίσης θέλουμε η νομική πράξη για την ε, γονική ευθύνη θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να υπάρχει η ισότητα μεταχείριση δανών και μη δανών υπηκών. Εγώ θα σταματήσω κύριε Πρόεδρε γιατί θα μπορούσα να μιλάω για πολλή ώρα ακόμη και θέλω να σας πω ότι Σήμερα μόλις έλαβα μια πάρα πολύ επικαιροποιημένη αναλυτική έκθεση, 200 περίπου σελίδες ε, από υπήκο της Δανίας. Δεν κατάφερα να ακόμη του συναδέλφου μου, θα το κάνω σύντομα όμω για αυτό το έγγραφο, αλλά καταλαβαίνετε, φαντάζομαι και εσεί, κυρία Πρόεδρε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουμε τι αναφέρουσε και τα παιδιά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βέρτμαν. Ποιο από τα μέλη τη ε, αντιπροσωπεία που βρίσκεται κοντά μα επιθυμεί. Α, καλά, μετά. Πρώτα λοιπόν το λόγο η κυρία Λου. Κομισιόν. Excuse me, if we are speaking... Θα πρέπει να απαντήσει η συνάδελφός μου που κάθεται εδώ δίπλα μου. Εσείς είστε η κυρία Χόφμαν. Εσείς. Ε, ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε θα μιλήσω από τη σκοπιά της ε, δικαστικής συνδρομής σε αστικά θέματα, σε αστικές υποθέσεις για απαγωγές παιδιών, για ε, κυδαιμονία κλπ. Ευχαριστεί η Κομισιόν την ε, Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής για τη χρήσιμη πρωτοβουλία που ανέλαβε για την βελτίωση των, δικαιωμάτων των παιδιών και των γονιών τους στη Δανία. Από την σκοπιά όμως του νομικού πλαισίου τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι ότι η Δανία χαίρει ιδιαίτερη θέσεως ό,τι αφορά τη δικαστική συνδρομή σε θέματα αστικού δικαίου, δυνάμει του πρωτοκόλου 22 της συνθήκης, η Δανία δεν συμμετέχει στη συνεργασία του κεφαλαίου 5 του τίτλου μάλλον 5 του κεφαλαίου 3 της συνθήκης, άρα δεν δεσμεύεται από την ενωσιακή νομοθεσία σε ό,τι αφορά απαγωγές παιδιών, κυδαιμονία και δικαιώματα επισκέψεως. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, σχετικοί κανονισμοί κλπ. Αλλά πρέπει να είναι σαφές το γεγονός ότι η νομοθεσία αυτή αναφέρεται μοναχά σε κοινού κανόνες δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτελέσεως των αποφάσεων σχετικά με περιπτώσεις απαγωγής παιδιών μεταξύ χώρων μελών και την άσκηση των δικαιωμάτων επισκέψεως. Όμως η χορήγηση του, δικαιωμά, του δικαιώματος προσβάσεως και, το, και η χορήγηση του δικαιώματος κυδαιμονίας δεν καλύπτονται από τον κανονισμό, αλλά παραμένουν στα χέρια των χωρών μελών. Εν πάση περιπτώσει, ο κανονισμός είναι όντως χρήσιμος για την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, περιπτώσεων απαγωγής παιδιών. Η Δανία, όπως και οι άλλες χώρες μέλη της Ένωσης, είναι συμβαλόμενο μέρος ε, στην συνθήκη του 1980 για απαγωγή παιδιών και επίσης στη συνθήκη 1966 για προστασία των παιδιών. Η συνθήκη του 80 καθιερώνει σύστημα συνεργασίας μεταξύ κεντρικών αρχών ούτω ώστε να διευκολυνθεί η αποκατάσταση επαφών για την επιστροφή στο status κουβό του παιδιού το οποίο απήχθη παράνομα, αφαιρέθηκε παράνομα από την ε, συνήθη κατοικία του. Ωστόσο, το σύστημα δεν επιτρέπει σε καμία αρχή να εποπτεύει το πώς εφαρμόζουν οι χώρες μέλη τη συνθήκη. Είναι σαφές ότι υπάρχει η Ειδική Επιτροπή της Χάγης η οποία συνέρχεται σε τακτά διαστήματα και δύο ειδικέ επιτροπές των συνθήκων του 1980 και του 1966 για απαγωγή παιδιών και προστασία παιδιών το 2011 και το 2012 όπου όλα τα συμβαλόμενα μέρη συζήτησαν το θέμα και προσπάθησαν να καταλήξουν σε κάποια χρήσιμη λύση. Ωστόσο δεν υπάρχει εποπτική αρχή δεν υπάρχει δηλαδή ένα είδος ευρωπαϊκού δικαστηρίου όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ένωσης. Αυτό είναι και το αδύναμο σημείο του συστήματος το οποίο συνδέεται με το γεγονός ότι η Δανία δεν δεσμεύεται από την ενωσιακή νομοθεσία για τη συνεργασία σε αστικά θέματα. Είναι λοιπόν σαφές ότι εδώ σημειώνονται κάποια προβλήματα. Τούτου λεχθέντους επιτρέψτε μου να δώσω να περάσω το μικρόφωνο στους ε, συναδέλφους μου της ε, Διεύθυνσης ε, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, εμείς εξετάζουμε κάθε περίπτωση που τίθεται υπόψη μας πολύ προσεκτικά για να δούμε εάν υπάρχει κάποια διασύνδεση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως είπα παρακολουθούμε την εξέλιξη των υποθέσεων για το μη νομοθετικό έργο και την ανταλλαγή πληροφοριών για τα δικαιώματα των παιδιών έχουμε μια ανεπίσημη εργασία για τα δικαιώματα των παιδιών όπου μπορούν και συζητούνται και στο μέλλον θα συζητούνται θέματα απαγωγής παιδιών έχουμε και το Annual European Forum για τα δικαιώματα των παιδιών που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβρη φέτος και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν εκεί είναι και η απαγωγή παιδιών από γονεί. Άρα τα έχουμε υπόψη όλα αυτά τα θέματα και τα παρακολουθούμε προσεκτικά. Σας ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Και ας ακούσουμε τώρα την κυρία Αούκεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα, δεν δήλωσα ότι τα δανέζικα δικαστήρια προβαίνουν σε διακριτική μεταχείριση. Εγώ ζήτησα μελέτη όλων των χωρών, όχι μόνο της Δανίας, για το εάν υπάρχει κάποια τάση να προτιμώνται οι πολίτες της συγκεκριμένης χώρας. Έχω την αίσθηση ότι ίσως αυτό να συμβαίνει. Ίσως όχι παντού. Γι' αυτό θα ήθελα να γίνει μια σχετική μελέτη. Γιατί βρίσκω ότι είναι ενδιαφέρον το θέμα αυτό για την ε, Επιτροπή Αναφορών. Όμως είναι λάθος να ακούει κανείς μόνο τη μία πλευρά σε μία περίπτωση διαζυγίου και να ακούγονται οι καταγγελίες της μιας πλευράς μόνο σαν να είναι δίθεν γεγονότα. Η αγαπημένη μου φίλη Αγγέλικα Βέρτμαν με την οποία συνεργάζομαι είπε κατά επανάληψη ότι αυτά είναι γεγονός γεγονότα δηλαδή, ότι ε, δηλαδή γίνεται κατάχρηση των δικαιωμάτων παιδιών. Όμως η ίδια η αναφορά λέει ότι πρόκειται για ισχυρισμούς. Άλλο ισχυρισμοί, άλλο γεγονότα. Αυτό που δεν κατανοώ Άλλωστε πολλοί από εμά θα έχουν ζήσει διαζύγια εδώ και γνωρίζουμε πόσο δραματικές μπορεί να είναι οι εξελίξεις και τι είδους ισχυρισμοί ακούγονται από τις δύο πλευρές ε, κατά της άλλης πλευράς κάθε φορά και δεν μπορώ να ψέξω τις δανέζικες αρχές ότι δεν μπορούν να συζητήσουν τις υποθέσεις διαζυγίων με τον τρόπο που τις συζητούμε εδώ. Άλλωστε, όπως είπα, δεν μπορεί να ακούσει κανείς μόνο τη μία πλευρά. Η αυστριακή υπόθεση Όλιβερ, που είναι πραγματικά ιδιαίτερα ατυχή υπόθεση, Όπω όμω λέει η αναφορά, υπάρχει απόφαση δανέζικου δικαστηρίου που δίνει την κυδαιμονία του παιδιού στον πατέρα. Αυτό όμω δεν αναφέρεται στην αναφορά. Γι' αυτό όμω οι δανέζικε αρχέ λένε ότι είναι απαγωγή ε, παιδιού. Εγώ δεν λέω ποιο έχει δίκιο, λέω μόνο ότι υπάρχει απόφαση από το 2010 του Δανέζικου Δικαστηρίου. Οι αυστριακές αρχές διαφωνούν, το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι Αυστριακό Δικαστήριο εξέδωσε άλλη απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε ποιο δικαστήριο έχει δίκιο. Είναι πολύ ατυχής περίπτωση όπως είπα πριν. Δεν νομίζω όμως ότι θα πρέπει ε, να εγκύψουμε τώρα στο πώς γίνονται, πώς προκύπτουν οι ισχυρισμοί στις περιπτώσεις διαζυγίου. Τώρα στη Δανία, οι πατεράδες δεν έχουν περισσότερα δικαιώματα από τις μανάδες. Έχουν μένει οι πατεράδες στη Δανία περισσότερα δικαιώματα από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εγώ χαίρομαι και είμαι υπερήφανο γι' αυτό, υπερήφανη γι' αυτό, διόλου δεν έχουν περισσότερα δικαιώματα από τι μητέρε. Είναι παράδοξο να ισχυρίζεται κανείς ότι οι πατέρες στη Δανία έχουν περισσότερα δικαιώματα από τις μητέρες. Εγώ πάντως το βλέπω αυτό. Η δανέζικη κυβέρνηση προσπάθησε να απαντήσει στις διάφορες ερωτήσεις μέσω της Δανικής αντιπροσωπείας εδώ στις Βρυξέλλες. Μπορεί οι απαντήσεις τους να μην είναι πλήρεις, ωστόσο ε, εγώ θεωρώ ότι προσπάθησαν να δώσουν ε, απαντήσεις και δεν νομίζω ότι οι δανέζικες αρχές θα μπορούσαν να είχαν ε, υπησέτηση στις λεπτομέρειες συγκεκριμένων υποθέσεων και ιδίως το ε, διαζυγίου. Και βέβαια ε, υποχρεώμαστε στη Δανία να, να συμμορφούμεθα με τις αποφάσεις των δικαστήριων και μπορεί άλλωστε να εφόσον αποδειχθεί ότι δεν εφαρμόζονται, δεν επιβάλλονται οι συνθήκες ή οι διατάξεις της συνθήκης, τότε κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι είναι ατυχές ότι η Δανία έχει επιλέξει να μην συμμετέχει, έχει, δηλαδή επιβάλλει έχει επιλέξει το opt-out από την συνθήκη αυτή. Και εγώ πάντως εργάζομαι υπέρ της άρσης του opt-out. Προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε παράλληλη συμφωνία αλλά μας το αρνήθηκαν. Ε, παράλληλη συμφωνία στο αστικό δίκαιο με την ε, συμφωνία για την κυδαιμονία των παιδιών, το ίδιο για τις πτωχεύσεις. Και εκεί μας αρνήθηκαν τη δυνατότητα να έχουμε ε, παράλληλη συμφωνία και βέβαια δεν μέμφω με τις άλλες χώρες με για παράλληλη συμφωνία, γιατί γνωρίζω ότι είναι μεγάλη φασαρία. Ωστόσο ζητήσαμε να διαθέτουμε παράλληλη συμφωνία και δεν μας δόθηκε η δυνατότητα. Και λυπούμε γι' αυτό πολύ, διότι όντως θίγονται και τα παιδιά και οι μητέρες και οι πατέρες και είναι πράγματι πάντοτε πολύ ατυχείς οι υποθέσεις αυτές. Όμως, επιμένω ότι πρέπει να γίνει μελέτη που ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου. Να εξεταστούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων στις χώρες μέλη για να δούμε αν κλείνουν υπέρ περισσότερο των ε, υπηκών των ε, οικείων χωρών μελών. Αγαπητή Μάργαρετ, μ' ακούς. Μ' ακούς αγαπητή Μάργαρετ. Δεν ξέρω αν η έκθεση πρέπει να γίνει να μην γίνει, κανένα πρόβλημα να γίνει. Μην ε, απατάσαι όμως. Δεν γίνεται παντού αυτό. Στη Δανία γίνεται. Και από εκεί έρχονται και οι αναφορές, γι' αυτό το λόγο. Αλλιώς θα είχαμε αναφορές και από άλλες χώρες, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία ήταν από εκεί. Και γι' αυτό πήγαμε στη Δανία. Γιατί οι αναφορές έρχονταν από τη χώρα σου, Μάργαρετ. Εγώ συμφωνώ με ένα πράγμα. Ε, από όσα είπες, ότι εσύ άκουσες μόνο τη μία πλευρά και όπως και στα διαζύγια πράγματι πρέπει να ακουστούν και οι δύο πλευρές. Αλλά εγώ έχω να πω και κάτι ακόμη αγαπητή μου Μάργαρετ Άουκεν. Είχε τη δυνατότητα κύριε Άουκεν να πά εκεί στην Κοπενχάγη και να δεις ε, πώς μας αντιμετώπισαν οι αρχές. Αλλά ούτε εσείς ούτε κανένας άλλος δεν ήθελε να είναι μαζί μας. Γιατί αν είχατε έρθει θα μπορούσατε ίσως ε, με την ομάδα σας να ε, ε πολλά από όσα ακούσατε εκεί. Αλλά είναι πολύ απλό να έρθεις εδώ να μας πεις ότι ναι, άκουσα μόνο τη μία πλευρά. Και ξέρεις ότι και σε πολλές άλλες ε, επισκέψεις που κάνουμε ακούμε τη μία πλευρά και περισσότερο. Αλλά εμείς πραγματικά ακούγοντας αυτά που μας έλεγαν μας σηκώνονταν η τρίχα. Και τι πρέπει να πούμε δηλαδή, ότι έτσι είναι η νομοθεσία. Είναι όπως λέμε στη χώρα μου, αν αρέσουν οι φακές της τρως, αλλιώς τις αφήνεις, έτσι είναι τα πράγματα. Και αν μας αρέσει ο νόμος ε, έχει καλό αν όχι δεν μπορούμε να παρέμβουμε στα προβλήματα ή στους νόμους της Δανίας. Και αυτά μας τα είπαν οι αρχές ε, της Δανίας, ε, με αυτά τα λόγια. Σε αυτούς που ήταν μαζί μου στην αποστολή αυτή, σε αυτό το ταξίδι. Δεν είναι λοιπόν θέμα ε, του δικαιώματος, ε, ότι οι καλύτεροι πατεράδες ή οι καλύτερες μητέρες, μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Μιλάμε για πατεράδες δανούς, αλλά οι μητέρες να είναι από τη Χοκόκ, τη Βόρεια Αμερική, την Ιταλία, την Νορβηγία κτλ. κτλ. Εκεί ήταν το θέμα. Και δεν ήταν θέμα ποιο έχει το πάνω χέρι ο πατέρα ή μητέρα, αλλά όπω είπε, δανεί πατεράδες απέναντι σε μητέρες από άλλες χώρες. Γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Αν ήταν μια δανή μητέρα που από έναν Ισλανδό, Νορβηγό, Ιταλό γονέα του απαγόρευε να δει ε, το παιδί, πάλι θα είχαμε πρόβλημα. Πάλι θα ε, διαμαρτυρόμαστε, όπως η κυρία Φέρτον που εξήγησε την κατάσταση πριν. Είναι λοιπόν κύριε Πρόεδρε νομίζω μια έκθεση για την ε, διερευνητική αυτή επίσκεψη που κάναμε στην Δανία. Θα έχουμε περισσότερες ε, ευκαιρίες να το συστήσουμε. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι μπορούμε να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Εγώ το έχω συζητήσει και με συναδέλφου, δεν ξέρω αν η κυρία Άουκεν ε, είναι διατεθειμένη να καλέσουμε εδώ τις ε, και αρχές. Πραγματικά να τις ξανακούσουμε τις ε, δανέζικες αρχές και να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψε για μια ακόμη φορά μαζί τους. Και να είσαστε εδώ παρόντες όλα τα μέλη της Επιτροπής Αναφών, γιατί πιστεύω ότι θα δείτε πού βρισκόμαστε. Ήδη έχουμε πάρει πάρα πολλές πληροφορίες, ξέρουμε πάρα πολύ περισσότερες λεπτομέρειε και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό και επιμένω να καλέσουμε τις δανέζικες αρχέ να έρθουν εδώ, μαζί και με τους αναφέροντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ο Γιάρ. Όπως είπαν και άλλοι, κάναμε την εξεταστική των πραγμάτων απόστολη, γιατί είχαμε τις σχετικέ σχετικές αναφορές μάλλον, και πήγαμε στην Κοπενχάγη, στη Δανία, χωρίς να θέλω να απευθύνω καμιά μομφή προς την Μάργαρετ την ίδια. Δεν πρόκειται για σένα μοναχά. Συνολικά πάντως εγώ δηλώνω ότι ευνηδιάστηκα. Συνήθως μετά από μια εξεταστική των πραγμάτων αποστολή λαμβάνουμε βοήθεια και από τους ε, άλλους βουλευτές από την ίδια τη χώρα στην οποία μεταβαίνουμε. Ούτε ένας δανός βουλευτής δεν ε, ήρθε μαζί μας ο οποίος να μπορούσε και να εξηγήσει λίγο την κατάσταση. Εκφράζω λοιπόν τη λύπη μου. Αντί λοιπόν fact-finding mission ήταν μάλλον μια φιλική περιφρόνηση. Ε, είχαμε πει τότε ε, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με τα αγγλικά. Δεν υπήρξε λοιπόν πραγματική κατανόηση. Το νιώσαμε και από την πλευρά των ίδιων των αρχών. Η Δανία θεωρεί ότι βρίσκεται στο δίκαιο της, δεν μετακινείται, έχουμε και τις αναφορές που μιλούν άλλη γλώσσα, δεν μπορούμε παρά να επαναλάβουμε μόνο τα όσα ακούσαμε και σημειώσαμε. Δεν είμαστε δικαστήριο, δεν μπορούμε να εκδώσουμε απόφαση, αλλά θεωρούμε καθήκον μας τα όσα ακούσαμε και ήταν και οδυνηρά πράγματα. Φτάσαμε μέχρι τα μεσάνυχτα σχεδόν με διαδικασία ακρόασης, όπως είπε και η κυρία Βέρθον, ο κύριος Σίτουργκάης, ε, και εγώ απαιτώ οι ερωτήσεις που έχουμε ακόμη να απαντηθούν από τις δανεικές αρχές. Και εκεί όπου είπαμε ότι έχουμε και πληροφορίες ποινικού χαρακτήρα. Θέλουμε να λάβουμε σχετική ενημέρωση και από τους ε, δανούς εισαγγελείς. Ακριβώς επειδή δεν είμαστε δικαστήριο. Τα κύρια προβλήματα για μας, διότι τα γνωρίζουμε και εμείς, έχουμε επισκεφθεί και ε, νεολαία κλπ. Και είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα Το πρώτο που μας ενδιέφερε πάντοτε, εάν η Δανία είναι τόσο πεπισμένη για το δίκαιο της νομοθεσίας της και θεωρεί ότι είναι και ο καλύτερος νόμος του κόσμου για, τα, για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, γιατί κάνει opt-out. Και εδώ είναι η πρώτη σύγκρουση. Αφενός έχουμε την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υποτίθεται δηλαδή ότι οι πολίτες της Ένωσης αναπτύσσουν ένα δικαίωμα, ένα σύνομο, ένα συνέστημα δικαίου και βλέπουμε, έχουμε αυτή τη τραγική υπόθεση από την Αυστρία, ότι εδώ πραγματικά αυτό δεν ισχύει. Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται έτσι Ευρωπαίοι πολίτες, ούτε μπορεί να διαμορφωθεί έτσι μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε και μια υπόθεση από την Πολωνία, τουλάχιστον εκεί λειτουργήσαν τα πράγματα. Βεβαίως όταν, όταν μαλώνουν δύο άνθρωποι πάντα υπάρχει πίκρα, αλλά τουλάχιστον μπορέσαμε να φτιάξουμε, να λειτουργήσει μια συνεργασία Γερμανίας-Ιταλίας. Και ε, λύθηκε η υπόθεση στο επίπεδο του ισχυόντος δικαίου. Δανία, όχι, κατεβάζει τα ρολά, λέει, δεν με ενδιαφέρει. Φτιάχνει στα γρήγορα μια δική της υπόθεση, μια δική της μάλλον απόφαση δικαστηρίου και αρκείται σε αυτά. Αυτό το opt-out με αυτή την περίφημη υποσημείωση κάποια στιγμή πρέπει να διαγραφεί. Δεν είναι πλέον επίκαιρη. Δεύτερη υπόθεση τώρα, πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή και θα ήθελα στην ακρόαση που διεξαγάγαμε να, είχαν, να ήταν παρόντες και δανείς συνάδελφοι. Ο καθένας βέβαια έχει τις ε, προσλαμβάνουσες παραστάσεις του, σε ό,τι αφορά και τραγικές περιπτώσεις ιδίω. Έχω μιλήσει και με ένα συνταξιούχο δικαστή νεότητας. Πρέπει το παιδί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η νέα νομοθεσία προβλέπει ωστόσο την υποχρέωση συνεργασίας μεταξύ των συζύγων. Αυτή η υποχρέωση συνεργασίας υποχρεώνει σε συνεργασία τους δύο ε, γονείς υπέρ του παιδιού. Αυτό όμως είναι και το ε, κέντρο των συγκρούσεων όταν πρόκειται για δανούς συζύγους. Διότι το παιχνίδι έχει την εξή εξέλιξη. Στη θεωρία, εντάξει, ναι, υποχρεωμένοι και οι δυο να συνεργαστούν, ε, πατέρα και μητέρα, δύο γονεί είναι όλοι και όλοι, που είναι αρμόδιοι, είναι υπεύθυνοι για το παιδί. Αυτοί καλούνται να συνεργαστούν. Ωραία. Μπορεί ε, να πάει προ το καλύτερο για τα συμφέροντα του παιδιού όταν συνεργαστούν. Στην θεωρία, στην πράξη όμως, όταν υπήρξαν περιστατικά, για παράδειγμα άσκησης βίας, που οδήγησαν και ε, στο διαζύγιο, αυτή η συνεργασία, η υποχρέωση της συνεργασίας είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η συνεργασία. Και εδώ, τώρα, ξαφνικά ο καλός γενικακός, κακός. Αυτός που δεν συνεργάζεται διότι λέει δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη μετά τα όσα έχουν συμβεί και που οδήγησαν στο διαζύγιο, δεν μπορώ να εμπιστευτώ το παιδί μου στον πρώην ε, σύζυγο. Άρα ξαφνικά εμφανίζεται ο, άλλος ε, ως μη διαθέσιμος προς συνεργασία και τότε αντιμετωπίζει τον νόμο. Το άλλο είναι, και είναι τμήμα του συστήματος, ορισμένοι πιστεύουν ότι η αγάπη γίνεται μίσος, συνεργασία τότε μισά-μισά εγώ έτσι τουλάχιστον κατανόησα, είναι πολύ περίεργη κατανομή, 3-2-4 μέσα στην ε, ε, εβδομάδα ή δεν ξέρω πώς, εάν ένας από τους δύο θέλει να πάει σε διακοπές, ας πούμε τρεις εβδομάδες, πρέπει να παρακαλέσει τον άλλο να το εγκρίνει πρώτα. Και αν ο ένας διαμένει στην Αμερική για παράδειγμα ή πάντως εκτός Δανίας, θα βγει ο άλλος και θα πει φοβούμαι ότι θα απαγάγει το παιδί. Να λοιπόν τώρα, και επομένω ο μη δανός σύζυγος έχει δεμένα τα χέρια του. Δεν μπορεί ποτέ να πάρει το παιδί να πάει να το ρίξει στου παππούδε, α πούμε ή σε άλλου συγγενεί. Έτσι λοιπόν το σύστημα οδηγεί τελικά στο αντίθετο αποτέλεσμα. Εγώ θα ήθελα, υποχρεώνομαι να το πω πολύ γενικά, να είχαμε δει έστω και κάποιες αρχές Μια διαφορετική συμπεριφορά των αρχών, να το πω έτσι. Δεν βλέπω ούτε καν ίχνος κατανόησης. Σαν να πέφτουμε σε ένα τείχο, όπως είπα προηγουμένως, μια φιλική περιφρόνησης. Εξηγήσαμε τον νόμο, είπαμε, μα ενδιαφέρει με νομοθεσία, αλλά εμείς ερχόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για αναφορές, για τις επιμέρους περιπτώσεις δηλαδή. Εμείς καλούμαστε να συζητήσουμε, όπως είπα, με μονομένες υποθέσεις, ατομικές υποθέσεις. Δεν χρειάζεται να έρθετε να μας εξηγήσετε το τι συμβαίνει ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και η Τουργκάης είπε σωστά. Αναμένουμε τώρα οι ερωτήσεις που έχουμε υποβάλει και που παραμένουν στο ακέραιο τους να απαντηθούν από τις αρχές. Και ίσως αυτές οι αρχές να δεχθούν τέλος πάντων να έρθουν και στην Επιτροπή Αναφορών για να συζητήσουν μαζί μας. Η κυρία Βέρτμαν έχει τελευταία το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη στην ανακεφαλαίωσή μου. Θα ήθελα να απευθυνθώ ε, στην Επιτροπή και να τους πω. Παρακαλώ να τοποθετηθείτε όσον αφορά την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και των κάθε μεμονωμένο αναφέροντα. Γιατί νομίζω ότι όλοι θέλουν να γνωρίζουν τις εξαιρέσεις σε σχέση με την Δανία. Και να πω στον Πίτερ ότι τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά, για όλα αυτά που είπε, με απόλυτη σαφήνεια. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να πω ότι μπορούμε να αντιδράσουμε και να αντιδρούμε γενικά μόνο με βάση αυτά που μας δίνουν οι αναφέροντες. Και σε αυτήν την έκθεση το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ε, καταγράφουμε τι ε, μαθαίνουμε, τι βλέπουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτα σαφές, κυρίως ε, για τους συναδέλφους, διότι δεν νομίζω ότι έχει σημασία και θα πρέπει να μας ρωτάτε τι πιστεύουμε και πώς αισθανόμαστε τότε δεν έχει νόημα. Τώρα, για τα στατιστικά δεδομένα. Σωστά είναι αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν στατιστικά δεδομένα, γιατί η διακριτική μεταχείριση δεν καταγράφεται ε, ως ε, τέτοια, άρα δηλαδή προφανώς εδώ υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, είπατε ότι δεν αναφέρατε κάτι τέτοιο και παραθέτω ότι πράγματι Υπάρχει κόκκος αλήθεια ε, σε αυτό που ισχύονται πολύ ότι οι Δανείοι προτιμούν να ευνοούν τους Δανούς γονείς. Επίσης, οι Δανείοι πράγματι ε, είναι υπέρ των Δανών σε μικτούς γάμους. Νομίζω λοιπόν ότι οι Δανείοι έχουν την άποψη ότι είναι καλύτερα για ένα παιδί ε, να μεγαλώνει στην ταινία. Αυτά τα λέω για να σας υπενθυμίζω. Και δεν είμαι και χαζή, τα λέω ε, για να τα θυμηθείτε όλοι. Όσον αφορά την περίπτωση της Αυστρίας, οι γονείς του Όλιβερ ποτέ δεν είχαν παντρευτεί και μετά θέλω να πω ότι είπε ο δικαστής ε, στις 21 Δεκεμβρίου του 2012 όπου ένας από τους τρεις δικαστές και υπήρχε και ένα τρίτο άτομο, δεν ξέρω πώς το πω στα αγγλικά, Υπήρχε λοιπόν ένας δικαστής με έναν εμπειρογνώμονα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγώ είπα ότι το παιδί αυτό έχει απαχθεί και αναφέρθηκα σε αυτό που είπε ο εμπειρογνώμονας γιατί είναι ένας ε, πραγματικά επαΐων για το θέμα αυτό. Να συνοψίσω αυτό που και ο Κάλλος θέλουμε μία επίσημη ακρόαση με εκπροσώπους, με υπουργούς, με αναφέροντες εδώ στις Βρυξέλλες για να καταλάβουμε τέλος πάντων τι γίνεται. Και για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους αναφέροντες και κυρίως τα παιδιά. Ευχαριστούμε την κυρία Βέρτμαν Κόλ. Κοίταξτε, Ναι. Να προσθέσω αυτό που λέει Ευαγγέλικα. Όχι, δεν σταμάτησα σε αυτό. Συνέχισα και είπα ότι αυτή είναι φαντάζομαι η κατάσταση στις άλλες χώρες. Ναι, το είπα εγώ. Και έχω ζητήσει να ε, δοθούν στατιστικά στοιχεία γι' αυτό, αλλά δεν υπάρχουν. Ή τέλο πάντων δεν έχουν. Φυσικά και δεν θα πω ότι είναι δυνατόν να είπα ποτέ ότι μόνο η Δανία έχει αυτό το θέμα αγγέλικα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, για τις παρεμβάσεις σας. Θα ξανακαλέσουμε τις ανέσικες αρχές. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση με την άλλη πλευρά. Προς το παρόν όμως δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ όλους. Κλείσαμε λοιπόν τις εργασίες μας για σήμερα γιατί το επόμενο θέμα για την υπηκότητα αυτό πρέπει να το αναβάλουμε γιατί ε, το όνομα του εισηγητή μου αναφέρθηκε σήμερα μόλις με email έτσι λοιπόν θα το συζητήσουμε αυτό στην ε, συναντήση των συντονιστών που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και παρακαλώ τους συντονιστές να μην απομακρυνθούν γιατί είμαστε στην ώρα μας για να ξεκινήσει η συνεδρίαση με τους συντονιστές.